Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Μερικές ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, οι διερμηνείς Σα με τα λύπη ότι συνεχίζεται η εργασιακή διαμάχη με τη δίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι συνθήκε εργασία που αποτέλεσε το αντικείμενο προειδοποίηση για περιακή κινητοποίηση. Η ποιότητα τη διερμηνία κινδυνεύει. Δυστυχώ λόγω τη διαμάχη αυτή η διερμηνία θα σταματήσει στι 6.30 όπω προβλέπει το πρόγραμμα τη συνεδρίαση. Και εμεί θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στο πώ θα χειριστούμε το πρόγραμμά μα για να μην βρεθούμε χωρί διερμηνία. Έχω και εγώ μια ανακοίνωση για την κοινή συνεδρίαση ΕΚΟΝΕΜΠΛ την 5η 28 Ιουνίου από τις 11 έως τις 12.30 με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης, τους ε, Επιτρόπους Μοσκοβισή και Τάισεν που θα ασχοληθούν με τις αναχώρες συστάσεις και ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στο σημείο 3, μία ανακοίνωση απλώς έχω για τον τελευταίο τριμερή διάλογο για την απόδοση έδρας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Ολοκληρώθηκαν οι σχετικές συζητήσεις σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα θέματα της ε, Τραπεζικής Αρχής, αλλά όχι ως προς το σκέλος των οριζόντιων θεμάτων. Και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και ο EMA και σε σχέση με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τι έντρε των οργανισμών. Η σχετική διαδικασία δεν έχει περατωθεί. Θα περιμένουμε λοιπόν νεότερα. Και τώρα περνάμε στο σημείο 4. Ήθελα να καλωσορίσω την ε, Μαργκρέτ Φεστάγκερ, την Επίτροπο επί του ανταγωνισμού. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο πρώτο μέρος του διαδρομένου διαλόγου μας για το 2018. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων που έχουν να κάνουν με τις δικές σας αρμοδιότητες σε βασικούς τομείς που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι θα σταθείτε στα πολύ σημαντικά ζητήματα της σωστής εξισορρόπησης μεταξύ των ε, κανόνων ανταγωνισμού και των ευρωπαϊκών εταιριών που θα μπορούσαν να ε, μας δείξουν και να φωτίσουν κάποιες ενδιαφέρουσες υποθέσεις, όπως την ε, κρατική φορολογία και ούτω καθεξής. Με αυτή την ανταλλαγή λοιπόν απόψεων, ήθελα να καλωσορίσουμε τη συμφωνία που πετύχαμε στον τριμερή διάλογο για το πολύ σημαντικό αυτό του ανταγωνισμού, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Μπορεί λοιπόν μια θετική απόφαση να είναι ε, χρήσιμη και σκόπιμη για να έχουμε ένα κατάλληλο δίκαιο ανταγωνισμού. Πρώτη περίπτωση συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου και ημών για την επίτευξη αποτελέσματος του τέτοιου στόχου. έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και πάνω απ' όλα τον Ραμόν Τρεμόζα, ο οποίος συνέταξε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση περί πολιτικής ανταγωνισμού που ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο. Ελπίζω ότι θα μπορέσω πολύ σύντομα να σας ενημερώσω για το πώς θα υλοποιήσουμε και θα δώσουμε συνέχεια σε πολύ συγκεκριμένα σημεία που ανέφερε η έκθεση. Αυτό που περισσότερο μου έκανε εντύπωση στην έκθεση ήταν η πρώτη παράγραφος όμως, η οποία λέει ότι οι επενδύσεις και η καινοτομία είναι καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Και νομίζω ότι έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ε, επενδύσεις και καινοτομία. Ο ανταγωνισμός και η επιβολή των κανόνων είναι το μόνο που μπορεί να μας βοηθήσει. Νομίζω όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να δούμε ε, την Ευρώπη να αναλαμβάνει πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο. Είναι όπως οι ποδοσφαιρικοί αγώνες. Ε, που όλοι προσπαθούμε να τους χωρέσουμε στο καθερινό μας πρόγραμμα αυτές τις μέρες. Αλλά αυτό ισχύει κυρίως για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να δούμε τους Ευρωπαίους πρωταθλητές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ανταγωνισμού με άλλες εταιρείε από άλλα μέρη του κόσμου. Το, οι ποδοσφαιρικές ομάδες και εταιρείε έχουν το εξή κοινό. Μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές μόνο εάν ε, οθηθούν να το κάνουν αυτό μέσω του ανταγωνισμού. Θέλουμε οι εταιρείε μας να επενδύουν και να καινοτομούν ε, για το μέλλον. Και θέλουμε αυτό να γίνει με όρους ανταγωνιστικούς σε ανοιχτές αγορές, διότι ο καλύτερος τρόπος να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές ε, για όποιον τον βρει θα πρέπει να αποτελέσει και αντικείμενο αμοιβή. Όσε εταιρείε λοιπόν είναι πρωταγωνίστριε θα πρέπει να μείνουν και στο διεθνέ προσκήνιο. Όχι αυτέ που δεσπόζουν επειδή ε, κατάφεραν να αυξήσουν ε, τα κέρδη του χάρη σε κρατικέ επιδοτήσει ή εξαγοράζοντα άλλε εταιρείε, εξαλείφοντα έτσι τον ανταγωνισμό. Οι εταιρείε χρειάζονται όμω και δυνατότητα ε, να έχουν διεξόδου σε σωστέ τιμέ και με τη σωστή ποιότητα. Γι' αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο ανταγωνισμό ε, υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της ε, αλυσίδας παραγωγής οξιών. Γι' αυτό θέλουμε να βρεθούμε στις διεθνείς αγορές με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν οι εταιρείε μας να ε, μπορούν να ανταγωνιστούν στις διεθνείς χρηματαγορές. Το Χάλιβας είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ε, χιλιάδες εταιρείε στην Ευρώπη με 30 εκατομμύρια εργαζομένους νομίζω περίπου εξαρτώνται από το Χάλιβα για την παραγωγή τους. Όταν λοιπόν η, Αρσερόλ, η Αρσελόρ Μιτάλ θέλει να αγοράσει την Ήλβα, τα μεγαλύτερα εργοστάσια χάλιβα στην Ευρώπη δηλαδή, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι τιμές του χάλιβα δεν θα αυξηθούν υπέρμετρα. Γι' αυτό εγκρίναμε τη συγχώνευση μόνον αφού η Αρσελόρ Μιτάλ ε, δέχτηκε να πωλήσει εργοστάσια σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιος που θέλει να συνεχίσει να λειτουργούν αυτά και να είναι ανταγωνιστικό στην ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να τα αναλάβει. Ο ανταγωνισμός οθεί τι επιχειρήσει να καινοτομούν. Όταν ισχυρέ εταιρείε ε, δεν μπαίνουν σε όρους ανταγωνισμού, μπορεί να πληγεί η καινοτομία. Γι' αυτό και οι προσφυγές μας κατά της Google πέρσι για ε, κατάχρηση της δύναμης που έχει η συσκευή αναζήτησης και την έλλειψη ευκαιριών για άλλους να ανταγωνιστούν ε, επί ίση όρη. Πάντως, η δουλειά μας στην, στην υπόθεση Google δεν ολοκληρώθηκε με την έκδοση της απόφασης μόνο. Θα πρέπει τώρα η Google να συμμορφωθεί με τον νόμο. Η ομάδα λοιπόν ασχολήθηκε ε, εντατικά με το όλο θέμα και μετά την απόφαση όπως και πριν. Η ουσία είναι ότι η Google θα πρέπει να έχει τους ίδιους όρους για τους ανταγωνιστές της όπως και για τον εαυτό της. Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν ανησυχίες για τους ε, αντιπάλους της Google που εμφανίζονται σε ένα κουτάκι για τις πωλήσει τους ε, στην αρχή της πρώτης σελίδας. Ξέρουμε ότι υπήρξε αύξηση στους αριθμούς αυτών των ε, εμπόρων, εμπορευομένων τους τελευταίους μήνες. Ε, μάλιστα τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ένας αντίπαλος της Google εμφανίζεται στο 1 τρίτο των παραθύρων της Google ε, σε σχέση με το 15% του περασμένου Μαρτίου. Δηλαδή αυξάνεται ο ρυθμός. Το ίδιο και ο ρυθμός των χτυπημάτων σε ε, πηγές πωλήσεων των αντιπάλων της αυξήθηκε από, σε 6,1% ε, από 1,5% το Φεβρουάριο. Αυτό για να γνωρίζετε πως έχουν ε, τα δεδομένα προ στιγμήν. Είναι πολύ νωρίς για να εξαγάγουμε ακόμη ακριβή συμπεράσματα. Επίσης συνεχίζουμε την ενεργό μας ε, παρακολούθηση και μιλάμε με τους συμμετέχοντες στην αγορά για να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τις απαραίτητες συνεισφορές για τη δουλειά μας και την παρακολούθηση. Το θέμα αυτό θα παραμείνει επιτάπητος και θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό. Θα παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα δηλαδή οι κανόνε μα για τι κρατικέ ε, βοήθειε, τι κρατικέ επιδοτήσει, που προσπαθούν επίση να οδηγήσουν σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Όταν οι πολυεθνικέ εταιρείε ε, ε, έχουν ευνοϊκή μεταχείριση ή τέλο πάντων επιλεκτικά τι μεταχειρίζονται κάποιε κυβερνήσει, όπω τα προνόμια τη φορολογία που δεν μπορεί να έχει κανεί άλλο, αυτό δυσκολεύει του μικρότερε καινοτόμε εταιρείε που πληρώνουν το δίκαιο μεριδιό του φόρου. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν επίση όρει. Άρα, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε αρκετές υποθέσεις ε, φορολογίας, κρατικής βοήθειας στην ουσία, με ειδική ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση και λάβαμε δράση για τις κατά των κατοχωρών για τη Fiat και την Amazon στο Λουξεμβούργο, για την στην Ιρλανδία και για 35 πολυεθνικές ε, στο Βέλγιο. Η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακόμη εξετάζουμε το τι συμβαίνει με τη McDonald's και την NGS στο Βέλγιο και κοιτάζουμε αν η IKEA έχει λάβει παράνομη βοήθεια στην Ολλανδία. Επίσης μας απασχολεί κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησαν τους κανόνες περί ξένων εταιριών εντός εισαγωγικών κανόνες που αποτελούν ότι πρέπει να παρεμποδίσουν την φοροδιαφυγή. Και κοιτάζουμε κατά πόσον έχει ευνοϊκή μεταχείριση κάποιες εταιρείε εις βάρος άλλων. Η ουσία είναι όμω ότι οι κανόνε για τι κρατικέ βοήθειε, τι κρατικέ επιδοτήσει ουσιαστικά ε, μπορούν να βοηθήσουν ε, στις επενδύσεις, επενδύσεις που τις χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη, επενδύσεις στις πράσινες υποδομές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα. Καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες μας επιτρέπουν αυτού του είδους τη ζωτική βοήθεια. Γι' αυτό συνεχίζουμε να ε, διευρύνουμε τον ε, κανονισμό μας περί μαζικών εξαιρέσεων. Να μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να δώσει μια βοήθεια χωρίς την έγκριση τη Επιτροπής εκ των προτέρων αρκεί να σέβεται τους κανόνες, τους σαφεί κανόνε που προστατεύουν τον ανταγωνισμό. Ε, κανόνες που ορίζουν ίσου όρου για όλου στην ε, Ένωση. Τώρα εξετάζουμε το πώς να ε, επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό μας για τι μαζικέ εξαιρέσει και να μπορούν οι κυβερνήσει να χρησιμοποιήσουν νέε ευκαιριέ που προτείνουμε για το ερχόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς ως Επιτροπή προτείνουμε ένα επενδυτικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αξιοποιήσει 15 δις από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να στηρίξει και να οδηγήσει σε 650 δις επενδύσεις. Το νέο πρόγραμμα επενδύσεων και έρευνας, ε, ορίζοντας Ευρώπη, με 100 δις ευρώ, ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε τόνο των επενδύσεων. Και τα δύο αυτά προγράμματα θα επιτρέψουν στα εθνικά κονδύλια να συνδυαστούν με ευρωπαϊκά και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το δυναμικό της Ευρώπης. Ο στόχος μας είναι να διευκολύνουμε όσο γίνεται τους ενδιαφερόμενους Ήδη έχουμε αναλάβει τα πρώτα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, όμως προτείνουμε το Συμβούλιο να διορθώσει τον σχετικό κανονισμό, ώστε να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε και τον κανονισμό για τις μερικές εξαιρέσεις. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει επίσης να εγκρίνει τη γνωμοδότησή του για την πρόταση αυτή, όσο το δυνατόν συντομότερα, ε, ώστε οι νέοι κανόνες περί ανταγωνισμού να αρχίσουν να ισχύουν εγκαίρως. Τώρα επεξεργαζόμαστε μια πρόταση για το πώς αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να διαμορφωθούν, αλλά το μόνο που μπορώ να πω προς στιγμή είναι ότι δεν πρέπει να είναι περίπλοκοι. Πολλές από τις βασικές αρχές των κρατικών βοηθειών ήδη είναι ενσωματωμένες στον ίδιο το σχεδιασμό των προγραμμάτων και πρόκειται για κανόνες όπως το αποφύγεται την απόθεση των ε, επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, αυτό δεν το θέλουμε, ή υποτροπή στην υπερεπένδυση, κατά τη υπερεπένδυσης. Διότι αν επενδύσουμε πάρα πολύ, κάποια πράγματα δεν θα γίνουν. Αυτές οι αρχές είναι ήδη ενσωματωμένες στα προγράμματα και αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε κανόνες που να είναι απλοί, ευέλικτοι. Και δύο τελευταίε κουβέντες για το Brexit. Ο λόγος για τον οποίο ε, είμαστε επιφυλακτικοί είναι γιατί δεν θέλουμε ο ανταγωνισμός να ε, πληγεί. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η δύναμη για, την, ε, για τις επενδύσεις, για την καινοτομία. Εάν κοιτάξετε τις οικονομίες μας, είναι τόσο στενά λένδετες που η κρατική βοήθεια που δίνει μια κυβέρνηση μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες στον ανταγωνισμό ανά την Ευρώπη. Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ένωση, ο δεσμός του με την, με την ε, ευρωπαϊκή οικονομία γίνεται λιγότερο στενός. Όμω, ακόμη και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν δίνει κρατικέ βοήθειε που υπονομεύουν του ίσου όρου για όλους. Γι' αυτό το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε κατευθυντήριε γραμμές για τις μελλοντικέ μα σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο και έχει αποδώσει ειδική προσοχή στον ανταγωνισμό και τι κρατικέ βοήθειε. Οι μελλοντικέ αυτές σχέσεις ε, απέχουν μόλις 10 μήνες στο μέλλον και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει κατεπηγόντως να κάνει επιλογές, να λάβει αποφάσεις και να υποβάλλει ρεαλιστικές προτάσεις για τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Η βασική πρόκληση εδώ για τις ερχόμενες διαπραγματεύσεις είναι πώς θα αποφύγουμε το σκληρό σύνορο, όπως εφαινομαστεί, στην Ιρλανδία. Για μένα, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την Ιρλανδία. Ε, αυτό ε, ούτω ή άλλω είναι σημαντικό από μόνο του. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η Ιρλανδία απομονωμένη. Είναι τα σύνορα τη ενιαία αγορά και τη Τελωνιακή Ένωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ακαιρεότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή. Και γιατί είναι αυτό σημαντικό. Δεν είναι επειδή ο ανταγωνισμό είναι αυταξία είναι γιατί ε, ο ανταγωνισμό μπορεί να μα προσφέρει ωφέλη σε όλου. Μπορεί να βοηθήσει τι εταιρείε και τι επιχειρήσει, του καταναλωτέ, να υποστηρίξει τι επενδύσει και την καινοτομία. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για όσα κάνετε και προσπαθείτε να τονώσετε τον ε, ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Είχαμε πολύ χειροπιαστά αποτελέσματα, συγκεκριμένα με τη Συμφωνία για την Ενδυνάμωση των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού, ώστε να μπορούν να αναλάβουν δράση και να προστατεύσουν τους καταναλωτές στην εθνική αγορά. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία σας και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι απτό σε σχέση με την καλή συνεργασία που μπορεί να έχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ευχαριστώ για τα λόγια σας και για την παρουσίασή σας και για όσα κάνετε. που υποστηρίζουμε ε, και εμείς σε αυτό το ζωτικό τομέα. Αναφέρατε την Google να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να πω και εγώ ότι ελπίζω το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί. Ως προς τον ανταγωνισμό, άλλωστε, απογοητεύτηκα όταν είδα ότι οι λεγόμενοι αλγόριθμοι του YouTube έδιναν ε, προτάσεις για βίντεο με πολιτικό περιεχόμενο σε μια στιγμή πολύ λεπτή για τα πολιτικά πράγματα της χώρας μου. Οι αλγόριθμοι του YouTube φαίνεται να είχαν σχέση με αυτό. Είμαστε ευάλωτοι και ευπαθείς εάν οι κανόνες δεν εφαρμόζονται με τρόπο υπεύθυνο από όλους. και διαδίδονται μέσω του διαδικτύου μηνύματα αποσταθεροποιητικά. Ο λόγος τώρα στους συναδέλφους, ο κύριος Χέις. Thank you, uh, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτροπέ Verstappen, Σα ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε και πάλι στην Επιτροπή μα. Σα ευχαριστούμε και για τη δουλειά που έχετε κάνει και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλα αναγνωρίση στην συζήτηση, στην Ελομέλεια, υποστήριξη της υποστήριξή σας για να υπάρχει μια εύρυθμα λειτουργούσα ενιαία αγορά, σε ό,τι αφορά και την πρόσβαση στην ενιαία αγορά, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολοι οι κανόνε ε, κατά καιρού για τα κράτη-μέλη. Δεν είναι το θέμα όμω αυτό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επαρκή ε, πολιτική ανταγωνισμού για να λειτουργεί η ενιαία αγορά για όλου. Μα υπενθυμίσατε και τέλο τη σημασία του Brexit. Ε, το καλωσορίζω αυτό και καλωσορίζω όχι μόνο τη σημασία τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τη σημασία να υπάρχει μια δίκαιη διευθέτηση του θέματο προκειμένου να μην υπάρχει αρνητική επίπτωση στι αγορέ, στι αμφότερε αγορέ και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, αυτά που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια, σε ό,τι αφορά τι καλύτερε επαφέ μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού. Τα καλωσορίζω λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία. Μία ερώτηση έχω να κάνω τώρα σε ό,τι αφορά μία ε, έρευνα η οποία ξεκίνησε από εσά το 2017 για την Ιρλανδία για, για ασφάλειες, ε, για οι κινητήρες στην Ιρλανδία σε ό,τι αφορά και τι συνθήκε που επικρατούν στην Ιρλανδία. Ξέρω ότι εσεί ξεκινήσατε την έρευνα αυτή και ότι έχει να κάνει με πρόσβαση σε δεδομένα, όπω για παράδειγμα ε, βαθμού πόντου ποινών κτλ. Κυρώσει που έχουν επιβληθεί και σε ό,τι αφορά την περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά. Μπορείτε να μα πείτε δύο λόγια για το πώ έχουν οι έρευνε. Είναι δύσκολο και πολύ σύνθετο προφανώ το θέμα αυτό και απαιτούνται πολλοί πόροι και από την ε, Γενική σα Διεύθυνση. Αλλά πότε περιμένετε κάποια πρώτα αποτελέσματα, κάποια προκαταρικά αποτελέσματα, γιατί ξέρω ότι πολλοί κόσμοι στην Ιρλανδία εξαρτάται από τη δουλειά που κάνετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό. Μια απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την εκτίμηση που εκφράζατε. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τις ανησυχίες στο θέμα των συνόρων και για τη σημασία εξέβρεσης απτών λεσέων για θέματα τα οποία θα επηρεάσουν και τον λαό της Ιρλανδίας αλλά και την υπόλοιπη Ένωση και ασφαλώς και τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα εκτιμώ το γεγονός ότι συμφωνούμε από αυτού. Σε ό,τι αφορά το το θέμα τώρα των ε, ασφαλίσεων για τα οχήματα, ξέρετε ότι έγιναν τον Ιούλιο του 2017 κάποιες επιθεωρήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη συλλογή πολλών δεδομένων Ετέθησαν κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια και κάποιες επερωτήσεις. Όταν ε, αναλύσαμε το σύνολο των απαντήσεων, θα αποφασίσουμε και για το επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Όπως είπατε, αυτό προφανώς και απασχολεί πολύ κόσμο και τους ασφαλιστές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιθετήσουμε το θέμα των συντομότερο Άλλη μια ερώτηση από αυτό. Στην παρούσα φάση θα μπορούσατε να μας πείτε, να μας δώσετε οποιαδήποτε ένδειξη για το πότε αναμένετε τα αποτελέσματα της έρευνας, γιατί καταλαβαίνετε λόγω της φύσης της έρευνας το θέμα αυτό απασχολεί πολλούς. Κατανοώ πλήρως, λέει η Επιτροπός Φερστάγκερ και γι' αυτό λυπάμαι ιδιαίτερος που δεν μπορώ να σας δώσω κάποιο χρονικό ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η φύση της έρευνα και θα πρέπει προφανώς να τηρηθούν όλοι οι κανόνες για σωστή διεκπαιρέωση. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα πρωτού ολοκληρωθεί η εργασία μας και θα πρέπει να γίνει σωστά η εργασία μας και καταλαβαίνουμε φυσικά α, πόσο σημαντική είναι η υπόθεση και του τουλεχθέντος θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να γίνει πιο γρήγορα η έρευνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Περέσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Μην νομίζετε ότι είμαστε λίγοι εδώ γιατί δεν ενδιαφερόμαστε για την πολιτική που ασκείτε. Όλοι γνωρίζουμε τη μεγάλη σας συνεισφορά για την επιτυχία του τελευταίου τριμερίου διαλόγου, ο οποίος καθόρισε πρότυπο υψηλού επίπεδου και αποτελεί υπόδειγμα και για τους επόμενους. Η Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι και η καλύτερη μέρα για τους συναδέλφους μου. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να σας θέσω τις εξής ερωτήσεις. Το γνωστό θέμα των McDonald's, το οποίο αναφέρατε έτσι επιγραμματικά, αλλά δεν μας είπατε και πολλά. Κάθε μέρα που περνάει, εμείς με το συνασπισμό των συνδικάτων που έχουν κινητοποιηθεί ιδιαιτέρως, ανακαλύπτουμε και νέες πτυχές αυτού του ζητήματος, οι οποίες έκδηλα μας οδηγούν στη σκέψη ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Όπως και να το ονομάσει κανείς και όπως και να το πει, Περί αυτού πρόκειται. Μιλούμε για εργασιακό dumping τελικά. Τι μπορείτε να μας πείτε για το πότε θα κλείσει η διερεύνηση της υπόθεσης και πού βρίσκεστε σε αυτό το θέμα. Και για τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές στο τραπεζικό τομέα, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, πώς αναλύετε τα τεκτενόμενα. Βλέπουμε ότι έχουμε νέο κύμα αναδιαρθρώσεων. Και τρίτο ερώτημα. σας δίνω μια ευκαιρία να ξεφύγετε από τη τεχνοκρατική ε, πτυχή που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρομαι στις πλατφόρμες. Η νομολογία ε, οδήγησε σε διάφορα νομοθετήματα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Με αυτά τα νομοθετήματα πιστεύετε ότι θα καλύψουμε όλα τα θέματα που θέλουμε να λύσουμε και κυρίως με αυτά αρκούν για να λύσουμε δύο ζητήματα που εμένα με ανησυχούν ιδιαιτέρως πρώτον ο σεβασμός της ιδιωτικής σφαίρας και ιδιωτικής ζωής από όλες αυτές τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές και δεύτερον η χρήση ε, που γίνεται σε αυτές τις πλατφόρμες για τη διάδοση των fake news, των ψευδών ειδήσεων όπως το ανέφερε και ο Πρόεδρός μας. Ευχαριστώ. Well, first of all, Καταρχάς, για τον τριμερή διάλογο, να σας πω ότι έχω μία νομοθετική πρόταση σε αυτή την ε, εντολή, σε αυτή τη θητεία και ήθελα να την αξιοποιήσω όσο το περισσότερο. Συμμετείχα σε όσους περισσότερους διαλόγους μπορούσα. Και η δουλειά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ε, έγινε και γι' αυτό ρήμασε το θέμα και μπορέσαμε να καταλήξουμε. Είναι μια σημαντική πρόταση. Χαίρομαι γι' αυτό. Τώρα για την υπόθεση των McDonald's. Όντω υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και δεν τι έχουμε όλες ε, ξεπεράσει. Προσπαθούμε να ε, τελειώσουμε τη δουλειά με τις διάφορες περιπτώσεις και ο όγκος της δουλειάς είναι πολύ μεγάλος. Για να μπορέσουμε να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές, χρειαζόμαστε περιστατικά, φακέλους, υποθέσεις και να ολοκληρώσουμε την εξέταση καθενός από αυτά. Ε, η υπόθεση με τα McDonald's θα είναι μία από αυτές τις υποθέσεις. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τώρα, για τον τραπεζικό τομέα. Δεν νομίζω ότι είναι οι αναδιαρθρώσεις αυτές καθ' αυτές που αποτελούν, που συνιστούν και την ύψιστη πρόκληση. Είχαμε κάποιες περιπτώσεις και τις έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, π.χ. τις δύο περιπτώσεις από την Ιταλία. Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Ο κλάδος αναπτύσσεται, υπάρχει fintech, Υπάρχει τεχνολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα, νέος τρόπος να γίνονται πληρωμές, νέος τρόπος να μεταφέρονται χρήματα και αναγκαστικά αυτό θα σπρώξει τον κλάδο να αναδιαρθρωθεί μόνος του. Ε, δεν έχω τα ισχυρά αριθμητικά στοιχεία, όμως ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τώρα από ό,τι ήταν ε, πριν από λίγα ε, χρόνια. Δεν αποκλείμε βέβαια το ενδεχόμενο κάποια τράπεζα να αντιμετωπίσει αρνητικέ εξελίξει. Όμω στο σύνολό του τραπεζικό τομέα είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι παλιότερα. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Όλοι ασκούμε πίεση για καλύτερε αγορέ κεφαλαίου, κεφαλαίου έτσι ώστε οι επιχειρήσει να έχουν πρόσβαση σε χρήματα και να μην οθούνται να πάνε στι τράπεζε και να δημιουργούν χρέη. Θέλουμε νέου επενδυτέ και ε, ε, νέες αρμοδιότητες στις επιχειρήσεις. Τώρα, οι ηλεκτρονικές και διαδικτυακές πλατφόρμες είναι ένα από τα πράγματα που με έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως. Και μένα και άλλους συναδέλφους. Εξημών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η κλάδη της οικονομίας ε, αναπτύσσονται διαφορετικά μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Οι δύο επιτροπές έχουν κάνει δύο διαφορετικές δημόσιες διαβουλεύσεις για να έχουν πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη με την πρόταση που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα οποία μας ήρθαν ως στροφοδότηση και συνεισφορά στη δημόσια διαβούλευση τα έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη οι επιχειρήσεις μας είπαν ότι κάποιος μας έκλεισε, μας πήγε τόσο χαμηλά ε, στο, ε, στην ε, σειρά εμφάνισης και ανάρτησης στο διαδικτύο που δεν είμαστε καθόλου ορατοί και δεν έχουμε καθόλου πελάτες. Έχει κάνει λοιπόν το δικαίωμα να ξέρει τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και σε ποιον θα πρέπει να στραφεί για να αλλάξει αυτό το τεκτενόμενο. Πρέπει να έχουμε νομοθεσία για κάτι το οποίο είναι προφανής επιχειρηματική πρακτική, ωστόσο πάρα πολλέ επιχειρήσεις ξανά και ξανά μας λένε ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και τους αφαιρεί κίνηση διαδικτυακή δεν έχουν και δεν ξέρουν σε ποιον να στραφούν για βοήθεια. Κάτι το θετικό ε, με αυτό το παρατηρητήριο είναι ότι είναι ένας πιο ευέλικτος τρόπος να εξεταστεί το θέμα με τις πλατφόρμες για να δράσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα αν προκύψει κάποιο ζήτημα. Και έτσι θα εξισορροπήσουμε, θα αντισταθμίσουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, Αντί να έχουμε νομοθεσία χωρί να ξέρουμε τι συγκεκριμένε επιπτώσει και άρα να έχουμε παχθεί και κοπιώδη γραφειοκρατική νομοθεσία, έχουμε παρατηρητήριο, το οποίο παρατηρεί τι συμβαίνει, βοηθάει την κατάσταση και αν τελικά αποδειχτεί απολύτω απαραίτητο θα έχουμε και νομοθεσία στη συνέχεια. Το σημαντικό είναι να ε, λειτουργήσουμε το συντομότερο, ε, όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Τώρα για τις ψευδείς ειδήσει, τα fake news δεν ε, αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου μου, αλλά με ενδιαφέρει ιδιαίτερο αυτό το θέμα. Όσοι νομίζουν ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, να ε, συνειδητοποιήσουν ότι κανείς δεν έχει ε, ε, εξετάσει την περίπτωσή τους αρκετά εξονυχιστικά προς το παρόν. Γιατί όλοι έχουν κάτι και είναι απολύτω δικαίωμά του. Κάποιος έχει μια ασθένεια, κάποιος έχει ένα διαζύγιο, κάποιος ο άλλος οτιδήποτε. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ιδιωτικής σφαίρας και δεν αφορούν κανέναν. Το σημαντικό είναι να έχουμε τους κανόνες να αρχίσουν να ισχύουν και το έχουμε από τα τέλη του περασμένου μήνα. Πρόκληση τώρα που αντιμετωπίζουμε είναι πια να τους εφαρμόσουμε, να τους υλοποιήσουμε, για να ξέρουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες πώς θα τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά. Αυτή είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση, να συνεργαστούμε, για να γνωρίζουν όλοι ότι μπορούν τώρα να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους. Συμμερίζομαι απολύτω τι ανησυχίε και του Προέδρου κ. Γκουαλτιέρη και τη δική σα κυρία Περβάν Μπερέ για τις ψευδείς ειδήσει, το σημαντικό είναι να έχουμε ενεργούς πολίτες, οι οποίοι να ασκούν κριτική σε οτιδήποτε τους παρουσιάζεται, επικοδομητική κριτική από με... Ε, σε οτιδήποτε τους παρουσιάζω εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε άλλος. Το καλύτερο οχύρωμα ενάντια στην προπαγάνδα και στις ψευδείς ειδήσει είναι ο ενημερωμένος ενεργός πολίτης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις τελευταίες ε, κουβέντες σας. Το εξετάσαμε, εξετάσαμε και τις απαντήσεις σας, τις ερωτήσεις αυτές. Ε, τις δημοσιεύσαμε. Δεν έχουμε λάβει απαντήσεις. Από το ECR δεν βλέπω κανέναν. Να περάσουμε λοιπόν στην άλλη, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τόρβαλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρα. Επίτροπε Βριστάγγεν, Λυπάμαι που καθυστέρησα. Unschoold και στα δανέζικα. Νομίζω ότι μετά τον πόλεμο στην Ευρώπη η καταπολέμηση των μονοπωλίων ε, και των ολιγοπωλίων ήταν υπερθμός ένα ε, πρωτεότητα. ο Κόντρα Αντενάουερ και στο πρώτο πρόγραμμα που κατάρτισε για το κόμμα των, Χριστιαν... δημοκρατών αυτό λοιπόν αποτέλεσε το πρώτο και πιο σημαντικό ζήτημα. Τώρα μιλάτε λοιπόν πλέον για πλατφόρμες, για ψηφιακές τεχνολογίες. Έχουμε πολλά πολυεθνικά ολιγοπόλια και μονοπόλια στην αγορά και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους με την Επιτροπή Τάξε για να τους βάλουμε σε τάξη κατά κάποιο τρόπο και αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα και σε πολλές εθνικές, ε, πολυεθνικές ευρωπαϊκές εταιρείες από ότι και σε άλλες. Ε, δεν θα βρούμε λοιπόν ε, λύση γιατί δεν θα πούνε οι Υπουργοί Οικονομικών ότι ναι πρέπει να σταματήσουμε. Όμως υπάρχει τρόπος να φορολογήσουμε τα μονοπόλια διότι αυτό θα γινόταν ένας πολύ χρήσιμος νέος ίδιος πόρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μπορεί να υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα μεν, αλλά είμαι σίγουρος ότι αν ψάξετε τα νομικά προβλήματα θα βρείτε κάποια διέξοδο και ως προς αυτό. Μιλάτε για κρατική βοήθεια. Ε, και το έχουμε ξανασυζητήσει σε αυτή την Επιτροπή. Εάν χαρίζουμε την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη σε ολιγάρχε ανά την Ευρώπη, δεν θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό ω παράνομη κρατική βοήθεια. Ευχαριστώ. Για την τελευταία ερώτηση. Νομίζω όχι. Εκεί βρισκόμαστε στα πολύ λεπτά όρια ...το τι μπορούν να συμπεριλαμβάνουν οι κανόνες κρατικής βοήθειας και τι μπορούν να πιάσουν ψαριά. Ε, δεν νομίζω ότι οι κανόνες κρατικής βοήθειας είναι σωστοί για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο που αναφέρεται, την πώληση της ιδιότητας του, Ευρω... του Ευρωπαίου πολίτη. Για τη φορολόγηση των μονοπωλίων. Το καλύτερο είναι να έχουμε ένα σύστημα φορολογικό που να λειτουργεί καλά Φυσικά και άκουσα και όλη την κριτική που ασκήθηκε για τις προτάσεις του Πιέρ Μοσκοβισή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των ψηφιακών εταιριών. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και κατεπήγον να ενημερώσουμε κάποιες βασικές έννοιες και το πώς ερμηνεύονται στην, ε, στη φορολόγηση των εταιριών. Αυτές οι βασικές λοιπόν ε, έννοιες είναι η δημιουργία αξίας και τι σημαίνει το να υπάρχει μόνιμο κατάστημα. Γιατί κάποιες από τις εμπορικές πρακτικές που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν είναι οι εξή ότι οι εταιρείε δημιουργούν αξία όχι με ε, έρευνα, και με προϊόντα, αλλά με τη συμπεριφορά των παρατών τους. Όπως για παράδειγμα εμείς ε, εδώ όλοι όταν κάνουμε μία αναζήτηση στο Google ε, χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη υπηρεσία και έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και ουσιαστικά δημιουργείται αξία χωρίς να υπάρχει καμία φυσική παρουσία στη χώρα μας στη χώρα αυτή που βρισκόμαστε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην όλη συζήτηση και προφανώς χρειάζεται ομοφωνία από πλευρά του Συμβουλίου για να ληφθούν αποφάσει. Άρα από το Κοινοβούλιο εξαρτάται να αναλάβει δράση. Γιατί αν δεν ενημερώσουμε κάποιε βασικέ έννοιε, τελικά θα καταλήξουμε σε, μια, σε ένα σενάριο όπου οι πολίτες θα χρηματοδοτούν το κοινωνικό κράτος, το κράτος πρόνοια. Τι βλέπουμε λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες εταιρείε και σε πιο παραδοσιακού κλάδους και βλέπουμε ότι μετά την πώληση και η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση για τη συντήρηση για παράδειγμα ενός προϊόντος, αυτό γίνεται σε ψηφιακό επίπεδο, το οποίο επίσης δημιουργεί αξία, παρόλο ότι το γεγονός ότι αποτελεί ψηφιακή υπηρεσία και μόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το πώς ε, εννοείται η δημιουργία αξίας όταν οι υπηρεσίες καθίστανται ψηφιακές και δεν σας λέω κάτι καινούριο, αλλά οι ψηφιακές εταιρείε πληρώνουν νέος 10, 9-10% φόρο επί της αξίας που δημιουργούν, ενώ άλλες εταιρείε πληρώνουν 23 24%. Δεν είναι δικαίως, λοιπόν ο ανταγωνισμός προφανώς και εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω τρεις ερωτήσεις για την Επίτροπο. Η πρώτη, που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, έχει να κάνει με την κατάκριση των βαθμολογιών, όπου υπήρξαν και ποινές από την Επιτροπή. Όμως σήμερα ρωτώ αν θα αναλάβετε κάποια δέσμευση εναντί των ε, πολιτών που έχουν πέσει θύματα απάτης και έστω και προκαταρκτικά να ε, εκδώσετε την απόφαση που έχει ληφθεί από το Δεκέμβριο του 2016. Είναι πολλές οι προσφυγές των πολιτών που έχουν μπλοκαριστεί και περιμένουν την έκδοση της απόφασης για την σχετική ε, κατάχρηση δεκαετία του 2000 από μεγάλες τράπεζες και τραπεζικούς ομέλους. Θέλω μια απάντηση γι' αυτό. Έπειτα υπήρξαν κάποια τυχή σχόλια στον τύπο πρόσφατα σε σχέση με τις πιέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εγκριθεί ε, το πανευρωπαϊκό συνταξιδοτικό προϊόν. Κάτι που θα επέτρεπε σε ορισμένους να βάλουν χέρι ε, σε μια πολύ ωραία σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς αξίας 2-3. Ε, Και τέλος, μια ερώτηση για τη διαχείριση των NPL. Ξε... Ήθελα να μου πείτε αν η γενική σας διεύθυνση ασχολείται με την δυνατότητα να αντιμετωπίσει ε, τα στρεπλωτικά αποτελέσματα στην αγορά από την αγορά και την κάλυψη των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εδώ κάποια κράτη έχουν δεχτεί βοήθεια ε, για να ξεπεράσουν αυτήν την κατάσταση. Άλλοι όχι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όλα αυτά ξεκινάνε και από την νομοθεσία και από την κεντρική τράπεζα. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί μια κατάσταση της αγοράς που διαρκώς πηγαίνει προς τα κάτω διότι όταν ε, κανείς οθείται να πουλήσει στην τιμή της αγοράς, τελικά η τιμή πέφτει. Ε, είναι και θέμα ανταγωνισμού. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε τη γνώμη σας σχετικά και αν υπάρχουν ε, έρευνες της Κομισιόν για το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτή την απόφαση, σε πολλές άλλες, υπάρχει δημοσίευση των αποφάσεων και μάλιστα τις τρομότερων δυνατόν. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει καθυστέρηση. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει το θέμα του απορρίτου των εμπιστευτικών πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση και σε περίπτωση αυτή υπάρχει μια ανταλλαγή επικοινωνία για το τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τι όχι. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι θεωρεί ο κόσμος ότι μπορούμε να μοιραστούμε. Όπως είπατε, Μπορεί να υπάρχουν ε, και ερωτήματα προς το δικαστήριο για ε, ζημίες σε προσωπικό επίπεδο και αυτό αποτελεί λοιπόν στόχο μας για κάθε απόφαση η οποία δημοσιοποιείται μόλις έχει ολοκληρωθεί η δικασία και δυστυχώ αυτό παίρνει κάποιο χρόνο σε ό,τι φορά τον BlackRock τώρα αν ε, ασκήθηκε πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το ξέρω. Αυτό δεν το γνωρίζω και ούτε είναι δικό μου θέμα το θέμα των πανευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών ταμείων. Υπάρχει φυσικά κρατική και από άλλα μέρη. Αυτό το γνωρίζω. Αλλά δεν γνωρίζω ποια ήταν η σχέση μεταξύ της BlackRock και των συναδέλφων μου. Σχόλια εκτό μικροφώνου για την τελευταία ερώτηση που κάνατε για τα, τα μη τα δάνεια. Το θέμα τη ε, πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει να κάνει με τι τιμέ τη αγορά και συχνά η τιμή τη αγορά είναι πολύ χαμηλότερη από την ε, καταχωρισμένη αξία. Αυτό σημαίνει προφανώ ότι θα πρέπει κανεί ε, να είναι σε θέση να τα πουλήσει και να πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει λοιπόν μια δευτερογενής αγορά για τα μη εξυπηρετούμενα δανεία, το οποίο θεωρώ ότι είναι ευπρόσδεκτο γιατί βοηθάει τα πράγματα. Γιατί αν ε, μπορεί κανείς να αγοράσει ένα τέτοιο δάνειο με 20 cents ε, και να το πουλήσει με 30, είναι καλή η υπόθεση. Φυσικά, αν δεν το καταφέρει αυτό, δημιουργείται ε, ένα δεύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες αποφάσεις που ελήφθησαν σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας για ρευστοποίηση, για να μπορούν να βγουν οι τράπεζες από την αγορά, από πλευρά ανταγωνισμού. Είναι σημαντικό αυτό. Οι τράπεζες οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά υποκαθεπτός πτώχευσης να μην συναγωνίζονται με πελάτες με τις άλλες υγιείς τράπεζες, να υπάρχει δυνατότητα ρευστοποίησης και να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά. Και έτσι απαλύνεται κάπω το βάρο από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τον Ιταλικό τραπεζικό κλάδο. Θεωρώ ότι η κατάσταση δεν είναι ακόμα ιδανική, αλλά είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Και σε ό,τι αφορά τη γενική εικόνα που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό φυσικά είναι στα χέρια του συναδέλφου του κ. Ντομπρόφσκη, αλλά και αυτό διαπιστώνει μια βελτίωση. Και είναι προφανώ επιβάρυνση για την ευρωπαϊκή οικονομία να υπάρχουν τόσα πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια θεωρώ ότι η τάση είναι θετική. Και φυσικά το γεγονός ότι δημιουργείται μια δευτερογενής αγορά είναι χρήσιμο για όλους. Ευχαριστώ κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο η οποία ήλθε σήμερα στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό κλάδο της βιομηχανίας που αναφέρεται και κάπως και στο θέμα της Google το οποίο αναφέρεται και σε ό,τι αφορά την όλη μεταρρύθμιση στο copyright. Μιλάμε για ψηφιακές, ε, παροχή ψηφιακής μουσικής. Η οδηγία για τα δικαιώματα, τα πραγματικά δικαιώματα, θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τις μουσικές πλατφόρμες on demand και από τα τέλη για άδειες που επιστρέφονται στον οικονομικό κλάδο. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό, ένα χάσμα σε αφορά την αξία αυτή και έχουμε και τη YouTube, μια εταιρεία η οποία κάνει web streaming σε 64% της αγοράς. Άρα έχει τεράστια συχνότητα πελετών. 600 εκατομμύρια πελάτες από 1,3 δις ε, παγκόσμιους χρήστες και 400 δις ε, δολάρια. Επιπλέον, η επιχείρηση αυτή εκμεταλλεύεται το δίκαιο για το copyright, το safe harbor θεωρεί ότι δεν είναι οι πλατφόρμες υπεύθυνε για την απόδοση των τελών στις, ε, στους ε, παραγωγούς. Ε, άλλες πλατφόρμες όπως το Spotify δεν αντιδρούν ανάλογα και πληρώνουν πολλά, για παράδειγμα, στους παραγωγούς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτές τις πλατφόρμες on demand, όπως είναι η YouTube, δεν πιστεύετε ότι πρέπει να εξετάσετε λίγο πιο επισταμένως τα πράγματα και το τι ισχύει η Επιτροπός. Όντως, το σκεπτικό σας είναι κάτι το οποίο έχει συζητήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν όχι απαραίτητα εγώ, αλλά οι συνάδελφοι. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να κλείσουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει, γιατί όπως είπατε κάποιες επιχειρήσεις φέρουν περιεχόμενο χωρίς να αμείβουν τους ε, παραγωγούς αλλά χρησιμοποιούν φυσικά για χρηματικούς σκοπούς την διάθεση του περιεχομένου για διαφημίσεις για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η πρόταση, αλλά ακολουθεί το ίδιο σκεπτικό ότι αν θέλετε να ωφεληθείτε από τις διαφημίσεις δίπλα στο περιεχόμενο, έχετε και κάποια ευθύνη για το ίδιο το περιεχόμενο και σημείο εκκίνησης, σημείο αφετηρίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ίδιο που ασπάζεστε κι εσείς, ότι θα πρέπει οι παραγωγοί κάπως να αμοιφθούν. δάλος θα σταματήσουν να παράγουν κάποια στιγμή. Και αυτό θα ήταν φυσικά επιζήμιο για όλους μας. Δεν ξέρω όμως πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η πρόταση. Ίσως να ξέρετε πολύ παραπάνω από ότι εγώ, αλλά σίγουρα ξεκινάμε από το ίδιο σημείο αφετηρία. Έχουμε και την δεύτερη φάση των ερευνών σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις. Κοιτάμε την ε, συγχωνεύση Apple με τη Shazam, ε. μια υπηρεσία αναγνώρισης μουσικής. Για να βρείτε το όνομα, για παράδειγμα, του καλλιτέχνη, η του τραγουδιού που ακούτε. Προσπαθούμε λοιπόν να διαπιστώσουμε κατά πόσον η απόκτηση της Αζάμ και τον, η προσάρτηση των κρατών της Σαζάμ θα επιτρέψει την προώθηση του Apple Music, τη μουσική τη Apple, σε βαθμό που θα βλάψει του άλλου παροχού. Δεν έχουμε ακόμα καθοριστική απάντηση, αλλά. Παρά το γεγονό ότι η Σαζάμ είναι μικρή επιχείρηση, αυτό που θέλουμε να καταλήξουμε και να αποφασίσουμε είναι τι θα γίνει όταν θα συμβεί αυτή η μεταφορά δεδομένων. και ελπίζουμε όταν τελικά ληφθεί η απόφαση να δημοσιευθεί επαρκώ και να κοινοποιηθεί επαρκώ για να το γνωρίσει όλο ο κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Ευχαριστώ Επίτροπε. Τρει ερωτήσει ε, έχω να κάνω. Καταρχά, ε, στην εισαγωγή σα είπατε για την ισορροπία μεταξύ ανταγωνισμού και των ε, Ευρωπαίων ηγετικών, ευρωπαϊκών ηγετικών επιχειρήσεων. Το θέμα λοιπόν είναι πώς ε, μπαίνουν όρια στην παγκόσμια αγορά και αντιμετωπίζουμε προβλήματα τέτοια και με την Κίνα και με, άλλους, ε, με άλλες χώρες που δημιουργούν πολλά προβλήματα στους Ευρωπαίους παραγωγούς και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε διατάξεις του 1989, απέρεψε διάφορα άλλα μέτρα σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο του Λονδίνου και του Βερολίνου ενέκρινε για παράδειγμα και άλλα συστήματα της Μοντσάντου, για παράδειγμα στο παρελθόν Ζήμες με πολιτική συμφωνία, ερωτώ, σε ό,τι αφορά τον τομέα των σιδηροδρομικών βαγονιών. Αυτό το θέμα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι αυξάνεται δραματικά ο παγκόσμιο ανταγωνισμός από πλευρά, από των Κινέζων. Δεύτερη ερώτηση, σε ό,τι αφορά το θέμα που μόλις αναφέρατε, σε ό,τι αφορά πολλούς μικρούς, ε, σε, σε ό,τι αφορά μικρούς παραγωγούς, μικρές εταιρείε, οι οποίες προσαρτώνται σε μεγάλες εταιρείε, όπως για παράδειγμα την Google. Πριν από κάποια χρόνια είχατε πει ότι η Facebook δεν είχε αγορά, δεν είχε αξία στην αγορά και ότι να ε, μας απασχολούσε. Σήμερα είναι μαζικά, μαζική εκμετάλλευση από τους δύο αυτούς ε, γίγαντες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιδρά. Δεν είναι, πιστεύω, σωστό αυτό. Τρίτη ερώτηση. Σε τι βαθμό η νέα κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου απέδωσε καρπούς. Πού πιστεύετε ότι εντοπίζονται τα περαιτέρω προβλήματα, γιατί αυτό μας απασχόλησε επισταμένως τα τελευταία χρόνια. Um, ναι, πρώτα απ' όλα για το θέμα των συγχωνεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποπτεύσει 3.000 συγχωνεύσεις τα τελευταία χρόνια. Το 5-6% εξ αυτών έχουν καθαριστεί, έχουν ρυθμιστεί, έχουν, έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή τους με διάφορα ε, μέτρα ε, έτσι ώστε να τηρείται το δίκαιο του ανταγωνισμού. Μιλούμε ε, πολύ για τι συγχωνεύσει όταν προκύπτουν ζητήματα, εκεί που ανακαλύπτουμε πράγματα. Και καλώ, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά το λέω για να έχετε και μια ιδέα από τις τάξεις μεγέθους. Τώρα για τις ζήμε και την Alstom. Προφανώ το τροχαίο υλικό και το υλικό σήμανσης και σηματοδότησης στους σιδηροδρόμους είναι ζωτική σημασία. Δεν είμαστε ασφαλείς αν δεν δουλεύει η σήμανση και η σηματοδότηση. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Επομένως θα εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτή τη συγχώνευση. Είναι σημαντικό ε, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να λειτουργούν τα πράγματα σωστά. Όλοι είμαστε υπέροχοι υπέρ του να μπορούν να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό ναι. Αλλά θέλουμε να έχουμε τη συνολική εικόνα της κατάστασης. Ποια είναι η πίεση ανταγωνιστική που υφίστανται από την Κίνα. Πώς οι κινέζικες επιχειρήσεις επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές και τις παγκόσμιες αγορές. Και θα αποκτήσουμε και την πλήρη εικόνα αυτό. Η συγχώνευση Siemens Alstom μας και γνωστοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου, είναι ακόμα πολύ νωρίς Εξελίσσεται η έρευνα, δεν έχω διαμορφώσει συγκεκριμένη άποψη ακόμα. Είναι δική μας υποχρέωση να μεριμνήσουμε, να κάνουμε το παν, έτσι ώστε αυτή η συγχώνευση, όπως και όποια άλλη συγχώνευση, γίνει με το σωστό τρόπο, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μην υποφέρουν από λιγότερο ανταγωνισμό ή από υψηλότερε τιμές. Αυτή είναι και δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αρμόδιας επιτρόπου της υποφαινόμενης. Εάν λοιπόν η έρευνά μας ε, αποκαλύψει ότι υπάρχουν ζητήματα ανταγωνισμού, τότε τα μέρη που συγχωνεύονται πρέπει να προτείνουν σχετικά μέτρα αποζημίωσης, εξισορρόπησης, αντιστάθμισης. Εμείς βλέπουμε όπου υπάρχουν επικαλύψεις όπου υπάρχουν ζητήματα υψηλού κινδύνου, όπου υπάρχουν θέματα διαχείρισης, τότε τα, τα μέρη πρέπει να προτείνουν τρόπους εξισορρόπησης. Θα επανέλθουμε όμως γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τώρα γιατί WhatsApp. Όταν την πήρε το Facebook, ήταν μικρή η εταιρεία. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησαν από την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα και γι' αυτό το κάναμε. Ερώτηση εκτό μικροφώνου. Απάντηση τη Επιτρόπου. Ένα από τα στοιχεία που εξετάσαμε ήταν ακριβώς το ζήτημα των δεδομένων. Τι θα γινόταν όταν η Facebook απόκτησε πρόσβαση στα δεδομένα της WhatsApp. Παρόλο που τότε είχε πει η Facebook ότι δεν θα συγχώνευε τα δύο σετ δεδομένων. Και ήταν πολύ καλό για τη Facebook που κάναμε ε, εμείς την ανάλυση αυτή, γιατί βγάλαμε τα αντίστοιχα πορίσματα. Μετά που οριστικοποιήθηκε η συγχώνευση, με την αλλαγή των ορών χρήσης ε, του Facebook, κατέστη εμφανές ότι θα μπορούσε η Facebook να συνδυάσει τα δύο σετ δεδομένων. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η συγχώνευση, αλλά το ότι δεν είχαν δώσει ε, όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις για αυτή την παράληψη ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμως έγινε μετά την ανάλυση που έδειξε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα ανταγωνισμού. Τελευταίο ερώτημα. Είναι πολύ νωρίς να ε, απαντήσουμε για το θέμα των εξουσιών των εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Έχουμε πολιτική συμφωνία, αλλά θα χρειαστεί κάποιος καιρός για να λυθούν τα νομικά ζητήματα, να πάρει νομική μορφή ο πολιτικός συμβιβασμός, να εγκριθεί στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και το Όμως, από τους συναδέλφους στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού του Ανταγωνισμού, όλοι αδημονούν να έχουν εργαλεία, διερευνητικά εργαλεία, να έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία, περισσότερους πόρους και μέσα για να κάνουν τη δουλειά και βεβαίως και τη δυνατότητα να επιβάλλουν κυρώσεις ύψους ικανού, ικανού ύψους ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζάνι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που βλέπω την Επίτροπο και τη διαθεσιμότητά της να μας απαντήσει στις ερωτήσεις μας να αναπτύξω λίγο ένα θέμα που με ανησυχεί εμένα και πολλούς άλλους. Μιλώ για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και την συνιστόσα τους που έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό όπου υπάρχει. Κατανοώ και θεωρώ ότι τα εμπορικά ζητήματα είναι κάπως εκτός του πεδίου αρμοδιότητάς σας, κυρία Επίτροπε. Ωστόσο, επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και ό,τι προβλέπουν αυτές. Άρα σας αφορά. Θέλω ε, να θέσω ένα ερώτημα για τις ΗΠΑ και να μας το σχολιάσετε. Όμως, προτού το κάνω αυτό, θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. Η, ε, η γεωργία και η παραγωγή αγροτικών προϊόντων την Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες ε, των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο με τις πρόσφατες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το ερώτημα, το ερώτημα πόσο τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα περιβαλλοντικά, τα εργασιακά, τα ποιοτικά, τα οικολογικά, τα περιβαλλοντικά και άλλα τηρούνται τελικά από τους εταίρους μας από τις τρίτες χώρες. έχουμε έλεγχο σε ό,τι αφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι τόσο μεγάλο έλεγχο όσο αφορά τους λοιπού. Όμω, αυτή τη στιγμή στι Ηνωμένε Πολιτείε ουσιαστικά διεξάγεται εμπορικό πόλεμο και ξεκινάει ένα τέτοιο εμπορικό πόλεμο. Καλωσορίζω τη βούληση της Ευρωπαίας Επιτρόπου να υπερασπιστεί και να ε, προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την ευρωπαϊκή οικονομία. Ποια είναι όμως τα συγκεκριμένα μέτρα που σχεδιάζετε να εθετήσετε κυρία Επίτροπε για να διαφυλάξετε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Πίτροπος, πράγματι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εκεί που υπάρχει ανησυχία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βγαίνει προς τα έξω, να ε, ε, μιλάει με διαφάνεια, να κάνει την επικοινωνία του, του, του περιεχομένου της εμπορικές συμφωνίες. Ο κύριος Χόγκαν και η κυρία Μάλστρομ είναι οι δύο αρμόδιοι επίτροποι για τις διαπραγματεύσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα μας στηρούνται και ότι δεν θα εισάγουμε αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ιδαλλιώς δεν θα είχαν γίνει ποτέ αποδεκτά. Ε, άρα, Σημαντικό είναι η επικοινωνία, την πρόσβαση που έχουμε στον κόσμο για να ξέρει ο κόσμος ποιο είναι το δυναμικό μιας συμφωνίας, ποιες δυνατότητες προβλέπει και προσφέρει. Νομίζω ότι η Σεσίλια κάνει αυτή τη δουλειά, Μάλστρομ, ε, για να μην φοβηθεί ο κόσμος. Θα ήταν κρίμα. Οι συγκεκριμένες εμπορικές συμφωνίες είναι μέρος της πολλά υποσχόμενης ε, διεθνούς εμπορικής ατζέντα. Δηλαδή, οι εμπορικές συμφωνίες τις οποίες συνάπτουμε τώρα έχουν ε, βάλει στο ντουλαπάκι της ιστορίας την έννοια του ελευθέρου εμπορίου. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε follower, να είμαστε ακόλουθοι. Θέλουμε να διαμορφώσουμε το εμπόριο. Το γεγονός ότι μπορούμε να ενώσουμε τον κόσμο, να καθίσει γύρω από, το, από ένα τραπέζι. Έχουμε οριστικοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, με την Ιαπωνία, με τη Σιγκαπούρη, τελειώνουμε με το Μεξικό, με τις χώρες της Νοτιού Αμερικής. Ξεκινούμε διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία και με την Αυστραλία. Όλα αυτά δείχνουν την εξουσία, την ισχύ, τη δύναμη της Ευρώπης, τη δυνατότητα της Ευρώπης να συγκεντρώνει ε, το κόσμο να τον συνενώνει όχι με το ελεύθερο εμπόριο της παλιάς σχολής αλλά με τη νέα ισορροπία του συσχετισμού των δυνάμεων που ε, είναι απαραίτητη. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται δασμούς για το χάλιβα και το ατσάλι και το αλουμίνιο στις Ηνωμένε Πολιτείες. Οι κύριοι Κατάινεν και Μάλστρομ, οι αρμόδιοι επίτροποι, ε, δουλεύουν πολύ επικοδομητικά για να ε, είναι προετοιμασμένοι να προσφέρουν την κατάλληλη απάντηση. Αυτό το είχα ξεκινήσει πρωτού προκύψει τέτοιο θέμα και τώρα βεβαίω είναι έτοιμη. Πηγαίνουμε στον ΠΟΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, γιατί μας χρειάζεται αυτό το πολυμερές νομικό πλαίσιο. Έχουμε επίσης μέτρα ε, αντιστάθμευσης, τα προϊόντα που αναφέρθηκαν και έχουμε και δικλείδες ασφαλείας και ρήτρες ασφαλείας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι οι δύο επίτροποι και έχουν την πλήρη στήριξη του σώματος των επιτρόπων, του συνόλου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι του στηρίζει και μα στηρίζει και το Συμβούλιο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν υποβάλει δασμούς, έχουν επιβάλει δασμούς και όλος ο κόσμο βλέπει ότι αυτό μα ενώνει. Γιατί επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο κάθε ευρωπαϊκή χώρα και η ισχύ μας ε, εξαρτάται από το βαθμό της ένωσης μας, έτσι ώστε να μιλούμε με μία φωνή. Thank you, Michael Raymond. Will be Ευχαριστούμε, κύριος Μία ερώτηση να κάνω στα γερμανικά, με επιτρέπετε. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο στην ομάδα εργασία ε, περί ανταγωνισμού έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από πλευρά τη Φρέντρικ Τζέινι από τον ΩΣΑ που εργάζεται στον τομέα του ανταγωνισμού εδώ και 10 χρόνια. Μας επεσήμαναν λοιπόν κάποια θέματα τα οποία ακόμα μα προβληματίζουν. Ε, δημιουργία και σχηματισμός τιμών από τράπεζε δεδομένων και επιρροή των τιμών από τράπεζε δεδομένων. Ε, έχουμε στον τομέα του ανταγωνισμού και σε άλλους τομείς μία μικροοικονομική αντίληψη ότι υπάρχει προσφορά και ζήτηση η οποία καθορίζει την τιμή και ότι όποιος ε, παρέχει μία υπηρεσία, ένα προϊόν, έχει λίγο πολύ την ίδια τιμή και σε ένα κατάλογο λίγο πολύ όλοι έχουν την ίδια τιμή. Αλλά δεν σημαίνει κάτι τέτοιο πλέον στο σύγχρονο εμπόριο online. Και αυτό λοιπόν επηρεάζει με πάρα πολύ μεγάλη τρόπο τις τιμές. Όποιος έχει καλύτερη τράπεζα δεδομένων μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες τιμές στους πελάτες τους και να διαμορφώσει έτσι την κατάσταση. Αυτό αλλάζει ή μπορεί να αλλάξει εντελώς την αντίληψή μας ε, περί αγορών σε ό,τι αφορά τις ε, online αγοραπολισίες και την εξέλιξη του τιμών. Όσα λοιπόν ε, κάνει σχετικές ε, έρευνες. Τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το παρακολουθεί το θέμα αυτό. Και πώς ε, μπορούμε ή πρέπει να αντιδράσουμε Μπορεί φυσικά να είναι πιο ευνοϊκέ οι τιμέ ε, για τον καταναλωτή, αλλά μπορεί να είναι και πιο υψηλέ η τελική ανάλυση βάσει τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται. Δεν μπορεί αυτό να το επιτρέψουμε να συμβεί. Δεύτερη ερώτηση, δεν είναι προ το συμφέρον μα. Δεύτερη ερώτηση, σε ό,τι αφορά την τελευταία έκθεση περί ανταγωνισμού και πάλι για την ψηφιακή αγορά. Το Κοινοβούλιο διαπίστωσε ότι στην περίπτωση τη εταιρεία Monsanto υπήρχαν και στοιχεία οικολογικά και δημοκρατικά τα οποία θα έπρεπε να λαμβάνονται πιο πολύ υπόψη σε ό,τι αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού στο μέλλον. Από πλευρά ε, δημοκρατία και πολιτική, πιστεύω ότι αυτό είναι ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το σχηματισμό τη ε, κοινή ε, γνώμη. Όταν μιλάμε για συγχωνεύσει, αλλά όταν μιλάμε και για κρατικέ επιδοτήσει, δεν μπορεί το μοναδικό κριτήριο στο μέλλον να είναι η λειτουργία τη αγορά. αν αυξάνεται η επιρροή της ε, Facebook και της ε, Google, ιδιαίτερα σε μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε, είναι προς το συμφέρον μας, να κοιτάξουμε κατά πόσον αυτές οι μεγάλες συγχωνεύσεις ε, θα επιτρέψουν τη διατήρηση μιας δημοκρατικής κατάσταση ενό δημοκρατικού καθεστώτος. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο την αγορά και τον ανταγωνισμό. Τι προτάσει λοιπόν θα προτείνετε, θα κάνετε για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του δικαίου περιεταγωνισμού. Απάντηση. Κατά πρώτον, χαίρομαι που θα είστε εισηγητής ε, της έκθεσης περιεταγωνισμού της επόμενης και που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και ευχαριστώ που αναφέρατε όσα κάνει η ομάδα του ΩΣΑ. Είναι πολύ σημαντικά, έχουν σοβαρή επίδραση και βαρύτητα, γιατί είναι πολύ καλά μελετημένα και είναι και ψηλή ποιότητα. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να μας εμπνεύσει και μας εμπνέει ήδη στη δουλειά που κάνουμε για την επιβολή του νόμου. Ένα από τα θετικά στοιχεία των πρόσφατων σκανδάλων είναι αυτή η ιστορία των υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν. Αυτό κατέρευσε και διαψεύστηκε. Ή πληρώνει με χρήματα ή πληρώνεις με δεδομένα. Και ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων θέλουν να πληρώνουν με χρήματα χωρί να χρειάζεται να θυσιάσουν τα δεδομένα του. Νομίζω στην Washington Post υπήρχε μια διαφήμιση που έλεγε ότι μπορούσε κανείς να δει και την τιμή των δεδομένων του την αξία όπου είχε κανείς ε, εναλλακτική είτε για περιορισμένη ε, πρόσβαση αλλά με τις διαφημίσεις και το tracking ενώ υπήρχε μια άλλη επιλογή, 50 δολάρια πιο ακριβή συνδρομή, όπου είχε κανείς πλήρη πρόσβαση, χωρίς κανένα tracking και καμία διαφήμιση. Αυτό δείχνει ότι μπορεί να βάλει κανείς ετικέτα με τιμή στα δεδομένα κάποιου. Δηλαδή, αντί να δίνει τα δεδομένα σου και να μπορεί κανεί να σου κάνει τάκι, να σε βρει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σου, γίνεται να πληρώσει παραπάνω και να μην συμβαίνει αυτό. Αυτό επιτρέπει στον κόσμο να έχουν μια πολύ καλύτερη αντίληψη του τι συμβαίνει. Και κάτι που αναφέραμε και προηγουμένως τα νέα δικαιώματα των πολιτών μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερο έλεγχο στα χέρια μας, να ξέρουμε ποιος μπορεί να δει τα δεδομένα μας και τι θα τα κάνει. Η ενίσχυση του αγωνισμού έχει ας πούμε να κάνει με το δικαίωμα στη φορητότητα. Μπορούμε να πάμε τα δεδομένα μας από τον ένα πάροχο να τα πάμε σε άλλο. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ανάδυση νέων υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τα μονοπόλια, δεν είναι απαγορευμένα τα πόλια βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού. Θέλουμε οι εταιρείε να μπορούν να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν. Όμω, αν κάποιο μεγαλώσει, αναπτυχθεί και γίνει δεσπόζων σε μια αγορά, τότε αποδυναμώνεται ο ανταγωνισμό. Έτσι λοιπόν έχει κανεί μια ιδιαίτερη ευθύνη να μην κάνει κατάχρηση τη εξουσία του για να ε, αμφισβητήσει τη θέση άλλων στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι δική μα ευθύνη να το διαφυλάξουμε αυτό. Να το βεβαιώσουμε. Και ω προ τα επιχειρησιακά μοντέλα και του τρόπου παραγωγή αξιών. Η παραγωγή αυτή καθεαυτή αλλάζει. Το κόστος μπορεί να περιοριστεί το κόστος του περιθωρίου και να φτάσει στα μηδενικά επίπεδα. Το θέμα είναι τι θέση μπορεί να έχει κάνει στην αγορά με τέτοιου είδους business model. Γι' αυτό έχουμε τρει ειδικού συμβούλου, του οποίου διόρισα φέτο και οι οποίοι ακριβώ θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Ελπίζω ότι όλοι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα. Ε, διάσκεψη θα έχουμε στις 17 Ιανουαρίου Και τελική έκθεση θα δημοσιευτεί του χρόνου την Άνοιξη. Για το παράδειγμα, της Μπάγερ και της Μονσάντο. ε, μπορεί να υπάρξουν θέματα ασφάλειας που θα ανακύψουν πέραν όλων των άλλων θέμα πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Είναι πολλά αυτά που μπορεί να προκύψουν όταν σχεδιάζεται μια συγχώνευση. Πρέπει να έχουμε όμως ειδικά εργαλεία για συγκεκριμένα θέματα. Στην συγχώνευση αυτή αγρογεωργικών χημικών που είδαμε φέτος, το θέμα είναι ποια είναι η θέση ακριβώ ε, των αγροτικών χημικών προϊόντων που έχει περάσει και έχει εγκριθεί και από αυτό το κοινοβούλιο. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στον τομέα αυτό και είναι πολύ δύσκολο μια εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στον τομέα. Είναι πολύ λοιπόν καλύτερο να λέμε ότι θέλουμε αυστηρού κανονισμού για το τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει παρά να περιμένουμε από το εργαλείο παρατηρήσεω των συγχωνεύσεων να ε, επιλύσει τις λεπτομέρειες ό,τι αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ε, αυστηρότερη προστασία του περιβάλλοντος αυτή εξ αρχή, αντί να περιμένουμε από την ε, συγχώνευση και το εργαλείο της να τα κάνει αυτά. Όσο για την κοινή γνώμη, μπορούμε να το δούμε από πολλές διαφορετικέ σκοπιέ. Σε ένα βαθμό οι κρατικές βοήθειε μπορεί να δώσουν δυνατότητα στο κοινό να διαμορφώσει άποψη, το είπαμε λόγου χάρη για τα μέσα που είναι ε, δημόσια. Μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά, αλλά να συνεχίσει να παρακολουθεί κανείς τις ειδήσει και από το feed του Facebook. Μπορεί κανείς να ε, αποφασίσει τι θα επιτρέπεται και τι όχι. Και η κοινή γνώμη να είναι πιο ποικίλη, πιο ενημερωμένη και να δούμε αν θα την την πραγματικότητα ή όχι. Τώρα για την παράνομη βοήθεια στα επιλεκτικά φορολογικά προνόμια σε κάποιες εταιρείε, αυτά σίγουρα επηρεάζουν και την ε, κοινή γνώμη που μπορεί να είναι πολύ αρνητική προς αυτό το είδος της βοήθειας. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε, κύριος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την ε, παρουσίασή σας. Μια γενική ερώτηση και μια ακόμη. Η πρώτη είναι πώς μπορούμε να δούμε τις συγχωνεύσεις. Διότι στα μικρότερα κράτη-μέλη έχουμε μεγάλους, ίσως και διεθνείς ανταγωνιστές που έχουν μεγάλη τάση προς τις συγχωνεύσεις. Οι προηγούμενοι επίτροποι κοίταζαν τις τοπικές αγορές Κάτι που ίσω επίπεδο ευρωπαϊκή αγορά να είναι καλό για να υπάρχει και αρκετό για να υπάρχει μια ισορροπία στην ευρωπαϊκή αγορά. Πώ αλλάζει λοιπόν η έμφαση από την τοπική αγορά στην ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια. Και μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για την Gazprom. Σημειώνω ότι υποχρεώσατε την Gazprom να τηρήσει κάποιες υποσχέσεις, κάποιες υποχρεώσεις δηλαδή να συμμορφούνται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και με κάποια πρόστιμα, ανάλογα με άλλων μεγάλων εταιριών, όπως η Apple, η Microsoft και ούτω καθεξής. Και επειδή ξέρουμε ότι η Gazprom οπωσδήποτε έχει υπονομεύσει τον ανταγωνισμό, όπως το είπατε και η ίδια, δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε αυτό. Όμως οι μεγάλες εταιρείες το κάνουν αυτό με την έλλειψη διαφάνειας, με πολιτικές πιέσεις και το καθεξής. Όμως, ξέρουμε ότι και για πολιτικούς λόγους η Gazprom έχουν ε, παρέμβει, παρέμβει και το έχουν μέσω αποδεχτεί. Πώς μπορείτε λοιπόν να χειριστείτε παρόμοιες υποθέσεις διαφορετικής εμβέλειας. Γιατί ας πούμε με το Nord Stream η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την άποψη το τοπίο και η αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού μπορεί να υπονομευτεί ή όχι. Για την πρώτη ερώτηση, πώς μπορεί κανείς να ε, εκτιμήσει την αγορά. Δεν αρκεί να βλέπουμε τι εθνικέ αγορές, συμφωνώ μαζί σα Πρέπει να βλέπουμε τι πραγματικέ αγορέ. Σε κάθε μια ξεχωριστή περίπτωση πρέπει να εκτιμούμε και να αποτιμούμε κατά πόσον υπάρχει κάποιο στον οποίο μπορούν να στραφούν οι πελάτε, καταναλωτέ. Διότι αν υπάρχουν νέε εταιρείε στι οποίε μπορούν να στραφούν οι καταναλωτέ, τότε υπάρχει ακόμη ανταγωνισμό. Αυτό που είδαμε τα τελευταία 5 έως 10 χρόνια είναι μισό της αγοράς να είναι εθνικό και το άλλο μισό να είναι ανοιχτότερο. Τώρα βλέπουμε το 65% όλων των αγορών να ε, έχουν ευρωπαϊκές διαστάσεις και μερικά να έχουν πάρει και παγκόσμιες προεκτάσεις. Οι εξελίξεις λοιπόν το πώς, του πώς βλέπουμε την αγορά, τις διάφορες αγορές, έχουν να κάνουν και με το πώς αντίνεται το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης Και οι περισσότερε εταιρείε ανταγωνίζονται και στο ε, διεθνές επίπεδο. Αυτά αντικατοπτρίζονται πολύ καλά στον τρόπο που κάνουμε την ε, ανάλυση μας της αγοράς. Πρόσφατα παραγγείλαμε και μελέτη για να δούμε αν οι κανόνες μας είναι στο ύψος, μάλλον στον ρυθμό των ε, τελευταίων εξελίξεων και κατά πόσο μπορούν οι εταιρείε μας να ακολουθήσουν τα επιχειρησιακά μοντέλα ως προς τα δάνεια, ναι, ήταν ε, όσο πιο καλά γινόταν προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα, ως προς την θέση της Κάσπρομ. Του στείλαμε μια δήλωση, μια αντίρρηση, όταν είπαμε ότι ε, η δήλωσή μας είναι ότι πιστεύουμε ότι κάνατε κάτι που ήταν αυτό, αλλά δεν λέμε ότι το κάνατε. Όταν προβλέπουμε υποχρεώσει για την Gazprom, ο στόχο είναι να πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είναι το θέμα να τηρούμε το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού μόνο. Υπάρχουν δύο πτυχέ. Και κάθε μια ξεχωριστά έχουν τη δυνατότητα, δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξη και ολοκλήρωση τη ευρωπαϊκή αγορά αερίου. Αυτό που είναι σημαντικό για κάποιον που αγορά, αγοράζει αέριο είναι να μπορεί να το ξαναπουλήσει. Το αγοράζει, πληρώνει θα πρέπει να μπορεί να το ξαναπουλήσει. Αυτό δεν συνέβαινε προηγουμένω λόγω συμβασιακών ε, περιορισμών. Δεν αρκεί όμω να αρθούν οι συμβασιακοί περιορισμοί. Πρέπει να μπορεί κανεί να το ε, παράσχει το αέριο, να το παραδώσει εκεί που θέλει να το παραδώσει. Εάν δεν μπορεί να πάρει πούμε, για να το πάει στου πελάτε του, πρέπει να μπορεί να έχει αγωγού αυτό ήταν το πρόβλημα με την Gazprom. Ε, ε, ότι πετύχαμε τελικά να μπορεί να ε, παρασκευτεί το αέριο εκεί που θέλουμε να παρασκευτεί. Ε, ας, πούμε, τη, ας δούμε τη Βουλγαρία. Η Gazprom τώρα υποχρεούται να προσφέρει αέριο και στις Βαλτικές και στη Βουλγαρία ακόμη και αν δεν υπάρχει δικό της, δικό της σύστημα αγωγών που να πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη σύμβαση και ε, στι βαλτικέ χώρε κάποιο Πολωνό, κάποια πολωνική εταιρεία θέλει να πάρει το αέριο και να το πάει στι βαλτικέ, αντί να το πάει στην Πολωνία, αυτό θα επιτρέψει να υπάρξει ασφάλεια στην παροχή και να αναπτυχθεί, να ανθίσει η αγορά του αερίου. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τι τιμέ, την τιμολόγηση. Δεν μπορούμε να ε, επιβάλλουμε μηχανισμού για τι τιμέ, εάν αυτό δεν γίνει μέσω υποχρεώσεων. Αυτό που υποχρεώνται τώρα να κάνει η Gazprom είναι να ξαναδεί τι τιμέ τη με μια θετική συγκριτική αξιολόγηση. κοιτάζοντα τι καθημερινέ τιμέ του αερίου στην Γερμανία και την Ολλανδία. Δηλαδή, εάν είναι συνδεδεμένε τι τιμέ του πετρελαίου, οι τιμέ του αερίου και ανεβαίνουν, θα πρέπει να ζητήσουμε ε, και να κοιτάξει κανείς να επιβάλλει και μια μείωση βάσει των πραγματικών τιμών στην αγορά. Αυτό είναι το σύνολο κανόνα που επιβάλλονται στην Κάσπρο. Αν δεν ακολουθήσουν τους κανόνες αυτούς θα επιβάλλουμε και πρόστιμα ή θα, ζητήσουμε, θα παρακύλουμε πλήρη έρευνα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι θα είχαμε πετύχει ε, υπό διαφορετικές συνθήκες. Ευχαριστούμε ο κύριος Χαουρέγγι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε και σας ευχαριστώ και για τη δουλειά που έχετε κάνει και για το ότι έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας να μας δείτε. Τρεις ερωτήσεις έχω να σας απευθύνω. Το μέρος του προϋπολογισμού που έχει προβλέψει η Επιτροπή για την αρμοδιότητά της. Operational expenditures, λειτουργικά έξοδα, λειτουργικές δαπάνες. Δεν έχω καταλάβει καλά τι είδου προγράμματα οικονομικά συγκεκριμένα θα χρηματοδοτήσετε. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα υποφεληθούν. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για αυτή την καινοτομία. Για το πόσο έχετε επιφέρει αυτές τις αλλαγές στον προϋπολογισμό. Δεύτερον, τραπεζική συγκέντρωση. στις διασυνοριακές περιοχές. Ουσιαστικά αυτό γίνεται παντού στην Ευρώπη και σε κάποιες περιοχές γίνεται ακόμα περισσότερο. Όμως έχουμε καταναλωτές, έχουν στεγαστικά δάνεια, έχουν επιστοτικές επεκτάσεις. Αναρωτιέμαι, βελτιώνεται η αγορά. Πολύ φοβάμαι ότι πόρο απέχουμε από αυτό. Και τρίτο ερώτημα, κυρία Πρόεδρε. η καταπολέμηση του αθέμητου ανταγωνισμού σε θέματα φορολογικά μεταξύ κρατών μελών. Δεν προχωρούμε όσο θα έπρεπε. Από τα σκάνδαλα του LuxLeaks μέχρι και σήμερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν υιοθετήσει ένα σωρό ε, ε, δράσεις για τα rulings, για τα tax rulings, τις ειδικές φορολογικές συμφωνίες μεταξύ κρατών και εταιριών, για τις διάφορες αποφάσεις. Ό,τι όμως και να κάνουμε, εγώ το μόνο που έχω καταλάβει είναι ότι ουσιαστικά αυξάνεται ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών. Έχουμε επαρκή μέσα για να ελέγχουμε αυτά τα κράτη και αυτόν τον έλεγχο να τον μπορούμε να τον κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχάς, να έχουμε ξεχωριστό προϋπολογισμό ε, ως Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό και την Ανταγωνιστικότητα είναι, ήταν κάτι το πρωτοφανές, το καινοτόμο, δεν το είχα ποτέ πριν και το θελήσαμε για να επενδύσουμε παραπάνω σε εργαλεία τεχνολογίας ε, ε, της πληροφορικής. Πρέπει να έχουμε, α πούμε, εργαλεία πληροφορική για να μπορούμε να βρούμε πράγματα που νόμιζε ο κόσμο ότι είχε διαγράψει και τελικά δεν έχουν διαγραφεί και έτσι ελέγχουμε του παρόχου. Έχουμε 800.000 έγγραφα. Για να μπορέσουμε να βρούμε ε, ε, ε, ε, εκεί, να πάρουμε μυρωδιά ε, του τι κάνει ένα καρτέλ, πρέπει να ψάξουμε 800.000 έγγραφα και πρέπει να, ε, πρέπει να έχουμε ένα εργαλείο πληροφορικής για να τα καταφέρουμε. Έχουμε αναθέσει μία μελέτη ε, σε μία εταιρεία για να μας δείξει πώς θα αξιοποιήσουμε τους αλγόριθμους στη δική μας δουλειά. για να δούμε τελικά με τον αλγοριθμό με ποιο ε, συνομωτεί κανείς ή με ποιον τα βρίσκει για να ε, λειτουργήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολλά εργαλεία πληροφορικής για να μπορούμε να κάνουμε τις σωστές έρευνες που κάνουμε στην αγορά. Πρέπει να μπορούμε να συλλέγουμε και τα στοιχεία και να κάνουμε έρευνα κλάδο. Μάθαμε πολλά από το κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, από την έρευνα για τις ε, ικανότητες και δυνατότητες αυτού του κλάδου. Από όλες αυτές τις έρευνες μάλθαμε πολλά και μας χρειάζεται προϋπολογισμός για να μπορούμε να τις διεξάγουμε και ενισχύουμε και τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Με την νέα νομοθεσία οι φιλοδοξίες μου πολλαπλασιάζονται. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα διάφορα εργαλεία που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να το κάνουμε. πιο, ο ξεχωριστό προπολογισμό. Τώρα για τη συγκέντρωση των τραπεζών δεν έχω πλήρη εικόνα. Ευχαριστώ να επανέλθω γραπτός και να σας πω τι έχουμε για τα θέματα Αυτά. Νομίζω ότι ο συνάδελφος Βάλτης Τομπρόφσκι είναι ο αρμόδιος επίτροπος. Με χαρά θα του το διαβιβάσω ότι ενδιαφέρεται η Επιτροπή σα για αυτό το θέμα. Το σημαντικό είναι ότι λειτουργεί αγορά και εξυπηρετούνται οι πελάτε. Βλέπουμε ότι επισέρχονται και νέοι παίκτε στον τραπεζικό τομέα και δίνουν νέου τρόπου πληρωμή και νέου τρόπου χρηματοδότηση. Προσφέρουν. Και τέλο, για το θέμα της καταπολέμησης του αθέμητου ανταγωνισμού και της παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Δεν έχει ακόμα κρυφθεί το κατά πόσο ήταν επιτυχημένη η δράση μας ή όχι, γιατί είχε ασκηθεί η προσφυγή και έκθεση εναντίον όλων των αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις. Ξεκινά τώρα η δευτεροβάθμια διαδικασία και στην περίπτωση της Fiat και στην περίπτωση της Starbucks. Το αποτέλεσμα θα το δούμε όταν αποφανθούν τα δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση η νομοθεσία που πέρασε στο Συμβούλιο ήταν πολύ σημαντική. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει κανείς να επενδύσει σε νέους ανθρώπους που μιλούν ξένες γλώσσες, που έχουν τις αρμοδιότητες, που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Όταν η νέα νομοθεσία αρχίσει να ισχύει, θα πρέπει να μπορούν όλοι να συνεργαστούν. Σε διάφορα κράτη-μέλη αλλάζουν την νομοθεσία. Δεν μπορεί να επαναληφθεί η περίπτωση της Fiat στο Λουξεμβούργο. Μία παρεμφερή υπόθεση δεν μπορεί να ξανασυμβεί στην Κύπρο. Στις κάτω χώρες άλλαξαν την νομοθεσία για, τις, ε, για τους συνεταιρισμούς και τώρα μόνο οι πραγματικοί συνεταιρισμοί ε, μπορούν να υποφεληθούν από αυτή την νομοθεσία στην Ιρλανδία έχουν τελειώσει αυτό με αυτό το ζήτημα του Double Irish. Τα κράτη-μέλη αλλάζουν την νομοθεσία και έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία που τίθεται σε ισχύ. Και παρόλο που αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μας για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Το Leaks και η δουλειά του Κοινοβουλίου ήταν πολύ σημαντική γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση και να επιφέρουμε τις αλλαγές που επιθυμούσαμε. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Η Εύα Μάιντεν παρακαλώ. Ευχαριστώ την ε, Επίτροπο για τη διαθεσιμότητά της και για τις ε, εμπεριστατωμένες απαντήσεις που μας δίνει. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω ε, ε, για την Gazprom. Είμαι από τη Βουλγαρία και για, διάφο... για πολλά χρόνια στη Βουλγαρία δεν είχαμε καμία ε, ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται με την Gazprom και τον αγωγό South Stream. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή απόφαση να έχουμε δεσμευτικές υποχρεώσεις και να υπάρχει νομική σαφήνεια. Ωστόσο, πολλοί θεώρησαν ότι παρέμενε ατιμόρυτη η Κάσπρο. Και πολλοί αναρωτιόντουσαν τι θα συμβεί εάν τελικά η Κάσπρομ δεν τηρήσει τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της. Γνωρίζω πολύ καλά τα πρόστιμα που θα μπορούσαν να επιβληθούν, τι θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει, θα χρησιμοποιήσει την εξουσία της για να ζητήσει πρόσβαση στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ζήτηση της Gazprom και των διαφόρων χωρών. Ευχαριστώ. Πέραν των όσων συζητήσαμε για την Gazprom και τις υποχρεώσεις της, το γεγονός ότι δεν μπορούν να ζητήσουν αποζημιώσεις για τον αγωγό South Stream που δεν ε, ε, ε, έγινε ποτέ, είναι σημαντικό. Ήταν σοβαρό το ποσό που συζητιόταν. Και θα ήταν μεγάλο βάρος για τη βουλγαρική οικονομία. το θέμα για μένα είναι ότι αυτή είναι η αρχή. Η αρχή επιβολής ενός νέου συνόλου κανόνων ώστε η Gazprom να δώσει τη δυνατότητα της θετικής ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς αερίου και θα υπάρξει και η ανάλογη ομάδα επενδυτών που θα κοιτάξουν εάν οι κανόνε τηρούνται. Το ίδιο και οι πελάτε τη Gazprom. Ελπίζουμε να μα ενημερώσουν αν δουν ότι κάτι δεν τηρείται. Εάν οι υποχρεώσεις ε, δεν γίνουν σεβαστέ, 10% του συνολικού κύκλου, είναι σημαντικό. Από τη στιγμή προβλέπονται δεσμευτικέ υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να γίνει έρευνα τώρα. Θα είναι πολύ πιο γρήγορη αντίδραση ε, εάν η Gazprom δεν ακολουθεί μη δεσμευτικέ υποχρεώσει. Αυτό είναι σημαντικό για να βεβαιωθούμε ότι Ακριβώς η απομόνωση της Βουλγαρίας και των ε, χωρών της Βαλτικής ό,τι φορά την παροχή αερίου θα πάψει και θα έχουμε και τις σωστές τιμές της αγοράς. Ακόμη και αν υπάρχει ε, η τιμαρρύθμιση με βάση το πετρέλαιο. Ευχαριστώ κύριε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. για τη δυνατότητα που έχουμε να θέξουμε κάποια ζητήματα. Θα μιλήσω και για τις ε, αεροπορικές εταιρείε. Γιατί γενικότερα ο κλάδος αυτός είναι από τους πιο κρίσιμους και τους πιο ανταγωνιστικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενιαία αγορά αεροπορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιφέρει τεράστιε αλλαγέ άλλωστε στον κλάδο. Σε ό,τι αφορά του διεθνεί ε, κανόνε, σε ό,τι αφορά του ευρωπαϊκού κανόνε. Έχει καταστήσει τι αεροπορικέ μεταφορέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο φθηνέ και πιο ασφαλεί και πιο προσβάσιμε ε, για όλου. Αλλά φυσικά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το έργο μα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μα για να υπάρξει πλήρη αξιοποίηση, πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού και για τις επιχειρήσεις και για τους επιβάτες. Υπολογίστηκε ότι μέχρι το 2035 η αεροπορική κίνηση θα αυξηθεί κατά 50%. Το οποίο είναι ένα ποσοστό απίστευτο σχεδόν. Αλλά προφανώ ο δίκαιο ανταγωνισμό είναι ακρογωνιαίο λήθο τη ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Γι' αυτό λοιπόν η οι παροχοί που παρέχουν ε, υπηρεσίες οι οποίες φαίνονται ανεξάρτητες ε, αποτελούν πρόβλημα. Για παράδειγμα, Lufthansa, Germanwings, ε, η Air France και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις που μας οδηγούν μοιραία στο ερώτημα κατά να αυτές οι μικρές επιχειρήσεις, ε, εταιρείε οδηγούν σε επιδείνωση και των ε, υπηρεσιών αλλά και των συνθήκων εργασίας σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική του ανταγωνισμού. Θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν πώς διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η συνεργασία μεταξύ παραδοσιακών αεροπορικών εταιρείων και φορέων ε, χαμηλού προπολογισμού δεν οδηγούν στρεβλώσεις. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, απαντάει η Επιτροπός. Γιατί ως τώρα αυτό που διαπιστώνουμε είναι πώς ε, μπορούν να συνεχωνευθούν ε, οι εταιρείε, οι αεροπορικές εταιρείε, προκειμένου να παρέχουν κοινέ όχι όμως με επίσημη σύγχρονευση για να μην υπάρχει θέμα μονοπωλίου, αλλά συνδυασμού τρομολογίων. Αυτό το θέμα όμω τη συνδιοκτησία μεταξύ του βασικού φορέα της βασικής ε, εταιρεία και της εταιρεία χαμηλού κόστου, πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι στην τομέα αρμοδιοτήτων μου, αλλά με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα το εξετάσω και θα σα ενημερώσουμε γιατί τα θέματα αυτά συγκέντρωση συντεκτησία και συντεκτησία είναι τα θέματα που μα απασχολούν στην παρούσα φάση να δούμε τι αποτέλεσμα υπάρχει όταν δεν υπάρχει επίσημα συγχώνευση, αλλά ουσιαστικά οι μέτοχοι είναι ίδιοι. Τι γίνεται λοιπόν με το, με το κίνητρο που έχει κανεί για να ανταγωνιστεί. Δεν έχω όμω αριθμητικά στοιχεία για να σας δώσω από πλευρά των αεροπορικών εταιριών. Άρα θα χρειαστεί να το μελετήσω και να σας ενημερώσω. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και λυπάμαι γιατί έχουμε και δύο συναδέλφου που είχαν ζητήσει το λόγο στην διαδικασία Catch the Eye, αλλά σα είπα ότι είναι πολύ αυστηρό το χρονοδιάγραμμά μα. Πόσο μάλλον που και οι διερμηνεί δεν μπορούν να παρατείνουν την περίοδο παροχή υπηρεσιών του έχουμε ήδη ξεπεράσει τον προβλεπόμενο χρόνο και θα πρέπει στο σημείο αυτό να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό την Επίτροπο Φερστάγκεν για την εξαιρετικά χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Πολύ, πολύ υποφελής και προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας. Ελπίζω να είναι εξίσου εξαίρετη. later. No, I think that So, let's move to next point of our. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της της διαταξής. Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ρέτζη. για την αύξηση του οικονομικού φάκελου για το, α, φάκελο, για το πρόγραμμα διαφορετικών μεταρρυθμίσεων από πλευράς ε, του Προεδρείου. Λοιπόν, εγώ είμαι εισηγητή και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του κοιόδη εισηγητέ και του συναδέλφου που κατέθεσαν 39 τροπολογίε. Δύο βασικά ζητήματα τα οποία και των οποίων άπτονται οι τροπολογίες, η γενική στόχοι του προγράμματος. Καταρχάς και ήδη όταν παρουσίασα το σχέδιο γνωμοδότησης είπα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει μια ευκαιρία να διευκρινιστεί και να διευρυνθεί η αντίληψη των μεταρρυθμίσεων για όλους τους τομείς. Συμπεριλαμβάνεται λοιπόν και ο τομέας βελτίωσης ε, της οικολογικής διάστασης των πολιτικών μας και της κοινωνικής συνοχή. Τα προγράμματα λοιπόν πρέπει να οδηγούν σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, σύγκληση και μία σειρά στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στο κείμενό μας. διάφορε τροπολογίες κατατέθηκαν από αυτού του θέματος και οι πιο πολλέ εξ αυτών έχουν τον ίδιο σκοπό. Παρουσιάζουμε λοιπόν συμβιβασμού για να δώσουμε μία απάντηση σε όποιο πολλές, όποιο πολλές γίνεται, σε όποιο πολλές τροπολογίες γίνεται από τις διάφορες ε, πολιτικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να τρέσουμε και μια αναλογία και μια ισορροπία μεταξύ των εκτιμώντας και του διακτατικού του κειμένου. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει λίγο πολύ με την χρηματοδότηση. Όλες αυτές ε, οι τροπολογίες έχουν να κάνουν με την εκ νέου χρήση των πόρων. αλλάζουμε λίγο τη διατύπωση, αλλά διατηρούμε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την έγκριση αυτή και θεωρώ ότι εδώ υπάρχει συμφωνία για την κινητοποίηση των ειδικών εργαλείων όπως προβλέπεται από το τρέχον MFF πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά λοιπόν συντομία για την ε, παρουσίασή μου και προσβλέπω στα δικά σας σχόλια, θα προσπαθήσω να τα λάβω υπόψη μου. Από την Ιβάνα Μάλετιτς, από ό,τι κατάλαβα, θα ακούσουμε την κυρία Σάντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της συναδέλφου Ιβάνα Μάλετικ που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Γι' αυτό και θα σας διαβάσω τα σχόλιά της στα αγγλικά. Εξετάζοντας τις τροπολογίες, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν υποβάλλουμε, δεν παρουσιάζουμε νέο κανονισμό για το πρόγραμμα στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο μετά το 2020. Το μόνο που κάνουμε είναι να αυξάνουμε τον προπολογισμό για το υφιστάμενο πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την χρονική περίοδο 2017 με 2020 κατά 8 ε, εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις ε, και όλες τις μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη με 222 εκατομμύρια ευρώ και γι' αυτό χρειάζεται η επιπρόσθετη δαπάνη των προγραμμάτων ε, των 80 εκατομμυρίων ευρώ διορθώνουμε Ενδεχομένως αυτό είναι άσκοπο. Είναι σημαντικό να μην προσδιορίζουμε τις μεταρρυθμίσεις εκ των προτέρων, διότι οι συνθήκες και οι περιστάσεις διαφέρουν από, το, από τη μία χώρα στην άλλη. Και αν θέσουμε προτεραιότητες με βάση τα συγκεκριμένα είδη μεταρρυθμίσεων, τότε τελικά ορισμένα κρατημέλη μπορούμε να τα περιορίσουμε, ίσως τα περιορίσουμε και δεν θα πρέπει να περιοριστούν να μην έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα. Τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη θα χάσουν ευκαιρίες αξιοποίησης του προγράμματος, διότι δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο και φορολογικό χώρο για αυτό το οποίο προτείνουμε ή γιατί έχουν καθορίσει διαφορετικές προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο. Η ιεράρχηση λοιπόν, η ιεράρχηση είναι κάτι το απαραίτητο λόγω των περιορισμών στον προϋπολογισμό και λόγω του υψηλού αριθμού των ετοιμάτων. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να λειτουργούμε με τη βάση προκαθορισμένων εκ των προτέρων μεταρρυθμίσεων, να έχουμε ε, μεταρρυθμίσεις με κριτήρια επιλογής που θα έχουν ιεραρχηθεί, που θα έχουν με επίπτωση συνέργειας ε, με άλλους κλάδες που θα αποσκοπούν στην οικονομική μεγέθυνση, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Απόψη μου είναι ότι ο γενικότερος στόχος του προγράμματος δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι γρήγορες αλλαγές. Ως Επιτροπή ΕΚΟΝ, Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, να τονίσουμε τη σημασία ε, που έχει όλα αυτά τα προγράμματα τελικά να προσφέρουν στήριξη στα κράτη-μέλη και στα κράτη-μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ, για να μπορέσουν αυτά να υιοθετήσουν τα κριτήρια και να συγκλίνουν το συντομότερο δυνατόν και στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα, με την υψηλότερη δυνατή κατάσταση. Άρα το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με την υλοποίηση και εφαρμογή των ειδικών συστάσεων αναχώρα που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, με δεδομένε τις προηγούμενε συζητήσει, είμαι βεβαία ότι θα συμφωνήσουμε πάνω στο περιεχόμενο αυτού του σχεδίου διατύπωσης και είναι σημαντικό να αναδείξουμε και να υπογραμμίσουμε ότι η αύξηση των κονδυλίων πρέπει να προέρχεται από το εργαλείο ευελιξίας Άλλωστε δεν είμαστε εμείς ε, υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Το ΕΣΥΑΡ δεν θα είναι παρέστα, εκπροσωπηθεί, άρα το λόγο έχει ο άλλος Τρεμόζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το ότι συμπεριέλαβε την προστασία μας σε ό,τι αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τι ευρωπαϊκέ μεταρρυθμίσει οι οποίε θα πρέπει να γίνουν σε αυτήν. Το ξέρετε και στην Επιτροπή αυτή. Συχνά έχω εκφράσει την άποψή μου αυτή. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί ένα θεσμικό όργανο το οποίο βασίζεται μόνο στο χρήμα. Έχει να κάνει και με τις βέλτιστες πρακτικέ. και υπό την έννοια αυτή θυμάμαι και την ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Ρίτα στο Τρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος και ανέφερε το Αμερικανικό Σύνταγμα. Όταν μιλάει λοιπόν για μια τέλεια ένωση, θεωρώ ότι στην όλη συζήτηση για το κατά πόσο χρειάζεται πιο πολύ ή πιο λίγη ένωση, θα πρέπει να μπει ο παράγοντας της καλύτερης ένωσης. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θεωρώ ότι είναι από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και δεν ξέρω κατά πόσον συμφωνείτε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή που συμπεριέλαβε την πρότασή μου αυτή. Ελπίζω δε. Να ρευθεί υπόψη αυτή η ιδέα και στο σύνολό της συγκλωματότησης. Αυτά. Ελπίζω επίσης να βοηθηθούν έτσι οι αθνικές κυβερνήσεις και υπηρεσίες να οργανωθούμε καλύτερο τρόπο και ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους κοιόδους. Ελπίζω να λεφθούν όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ποιος θέλει το λόγο. Μάρλε, θες να πάρεις το λόγο για τον Φίλιπ. Όχι. Ούτε και από την Γκουε βλέπω κανέναν. Ούτε από το EFTD, ούτε από το ENF. Κάτσε the έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και θα μας, ε, πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη επιτυχία ε, ακολουθείτε το θέμα αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρουσες ε, συμβαστικές σας προτάσεις. Να πω δύο λόγια για αυτά που είπε ο συνάδελφος από το ΕΛΚΑ, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα απευθύνεται σε όλα τα ζητήματα, αλλά με τα λίγα χρήματα που έχουμε και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει για να δώσουμε στους πολίτες μας αυτά που έχουμε υπόσχεθεί και να μην δημιουργούμε ε, τη μία απογοήτευση μετά την άλλη σε ό,τι άλλο, σε αφορά λοιπόν τους συμβιβασμού. Πιστεύω ότι δεν ήταν λάθος ε, μήνυμα. Όλοι χαίρονται για την... Ε, όλοι μάλλον χάρηκαν την προηγούμενο έτος με την έγκριση του κοινωνικού πυλώνα. Τώρα που πρέπει όμως ε, να υλοποιήσουμε την αρχή αυτή με τα προγράμματα αυτά, προφανώς υπάρχουν και δραστατικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα υλοποιήσουν το κοινωνικό πυλώνα. Δεν καταφέρνουμε όμως τώρα πλέον να συμφωνήσουμε. Είναι λυπηρό. Κρίμα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. στις αιτιολογικές σκέψεις έγινε μία αναφορά η οποία όμως δεν θα περιληφθεί στα άρθρα. Θεωρώ ότι έτσι και το μήνυμα αποφέρεται. Στις αιτιολογικές σκέψεις δεν περιλαμβάνεται, ναι. Το κείμενο φυσικά θα το μοιράσουμε. Μιλάμε για να χρηματοδοτήσει για ένα στενό χρονικό περιθώριο και μετά θα έρθει το καινούργιο πρόγραμμα στο οποίο θα είμαστε και η καθήλια αρμόδια επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό έχει αποφασιστεί πλέον και έτσι θα έχουμε δυνατότητα να δημορφώσουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο με πιο πολλούς πόρους, ελπίζω, για να συζητήσουμε πιο εκτεταμένα τα πράγματα αυτά, γιατί στα πλαίσια μια γνωματότηση τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα και έτσι δεν μπορεί να τεθεί πλήρω το θέμα τη αναχρηματοδότηση. Αναφέρεται στι ιδεολογικέ σκέψει ο κοινωνικό πυλώνα. Σα ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τη συνεργασία. Αύριο θα ψηφίσουμε και τις συμβαστικές προτάσεις θα τις λάβετε πριν από τη συνάντηση πριν από τη συνεδρίαση. Θα ψηφίσουμε και έχουμε πολλές ψηφοφορίες αύριο. Και μπορούμε λοιπόν στο σημείο να ολοκληρώσουμε και να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Να ευχαριστήσω τον Λούτο, ο οποίο θα αναλάβει και την Προεδρία. downgrade myself a little bit. Uh, so, we have... Μάλιστα, έχουμε το σημείο 6 στην ημερήσια κατάξη, τροποποιημένη πρόταση για τα μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ο κύριος Τσίλε είναι ο εισηγητής μας, ο οποίος δεν είναι και εδώ. Δεν είναι παρόν. Έχει αποστέλει ένα σημείο το οποίο και θα διαβάσω αξιωματό του. εσύ εισηγητή θα ήθελα καταρχά να ζητήσει συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ όλε τι ομάδε και του σκιώδει εισηγητέ του για τι συνεισφορέ του και για την συζήτηση που θα έχουμε σήμερα. Ο εισηγητή συμμερίζεται την άποψη ότι η διασυνοριακή φορολογική απάτη είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Το σημερινό σύστημα εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει του αυξημένου ρυθμού των οικονομικών συναλλαγών. Γι' αυτό φοβάται ο εισηγητή ότι ο φάκελο για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ πρέπει να εγκριθεί ω τα δυνατόν συντομότερα. Και αυτό για να δούμε την ε, τον αυξημένο όγκο χρηματοοικονομικών συνελλαγών. Οι αναφορές αυτές είναι σημαντικές και ο εισηγητής σκοπεύει να κάνει τις ανάλογες τροπολογίες. Στο πνεύμα κάποιων συμβιβαστικών λύσεων, ένα, μάλλον δύο ή περισσότερα κάτι μέλη μπορούν να ζητήσουν κάποια έρευνα σε σχέση με τα θέματα απάτης του ΦΠΑ. Επίσης, ο εισηγητής βάσει των τροπολογιών πιστεύω ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχουν μείζονες διαφωνίες. Γι' αυτό ο εισηγητής πιστεύει ότι αύριο στην ώρα των ψηφοφοριών θα πετέχουν θετικά αποτελέσματα. Αυτά από τον εισηγητή. Να ρωτήσω ποιο θα εκπροσωπήσει του Σκιώδη. Ο Μπράιαν Χέι. Βλέπω ότι αντικαθιστά τον κύριο Μάτο εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Προσωπικό εκ μέρου του κυρίου Μάτο του συναδέλφου μου να ζητήσω συγγνώμη, δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Συμμετέχει σε αντιπροσωπεία του ΕΛΚ για τις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία και την, την παρατήρησή τους. Συμφωνεί με την αποτίμηση του συγγητή ότι οι συμβαστικές λύσεις προτείνουν ένα καλό ε, σκόπιμο αποτέλεσμα. Και μου ζήτησε να αναφέρω τα εξή. Σαφώς τα τελευταία χρόνια το σύστημα ΦΠΑ δεν έχει παρακολουθήσει τους ρυθμούς εξέλιξης της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης όλων των οικονομιών μας και το τεράστιο ζήτημα που αυτό ε, δημιουργεί για το σύστημα ΦΠΑ και όλο το φρολικό κώδικα. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όλο σύστημα για την φορολόγηση του εμπορίου μεταξύ των κρατών είναι προσωρινέ διευθυντήσει. Ο ΦΠΑ είναι μια αυξανόμενη πηγή φορολογικού εισοδήματο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για τη σωστή κατανομή των φορολογικών εισόδων μεταξύ των 100 μελών, θα υποβάλουμε τη σωστή, την ονείλογη τροπολογία αύριο. μάλλον ελπίζουμε η τροπολογία που υποβάλλει σχετικά να το ψηφιστεί αύριο, όπω ε, όπως την υπέβαλε ο κύριο ΜΑΤΟ, για να ε, παραμείνει ο ΦΠΑ αυτή η σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων. Ο κ. Μάτο ευχαριστεί όλου του σκιώδει και τον καθένα αρμόδιο συγκητή για την αρμονική συνεργασία που είχαν και τη διάθεση να βρούμε συμβασμού. Πρέπει να αποστείλουμε στο Συμβούλιο το μήνυμα ότι θέλουμε περαιτέρω διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα ζωτική σημασία για τη φορολογία ω Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ευχαριστούμε κύριε Χέι. Έχουμε τον κύριο Λούτβιξον από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή, τον κύριο Τζίλε, για την πολύ καλή συνεργασία. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα οριστικό σύστημα, ένα νέο σύστημα ε, ΦΠΑ, διασυνοριακό για να φορολογείται και το σχετικό εμπόριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει την καλύτερη συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοικητικών αρχών των κατομελών. Πολλά χάνονται λόγω της έλλειψης επαρκούς συνεργασίας. Είναι λοιπόν πολύ καλό και θετικό αυτό. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να πάνε στον τομέα υγείας μας, ε, στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, Επίσης συμφωνώ με τον εισηγητή στην ιδέα του ε, φορολογούμενου ε, να μπορούν οι αρχές εύκολα να ελέγξουν τις εταιρείε για να είναι βέβαιες ότι δεν πρόκειται για περιπτώσεις προσπάθειας απάτης ή για τις περιπτώσεις της απάτης καρουζέλα, ας πούμε, που θα πρέπει να μπορούν να ερευνήσουν εύκολα. Επίσης, θα πρέπει να είναι δυνατό για τις φορολογικές αρχές να διεξαγάγουν έρευνες και σε αλλα κρατημέλη, Το τωρινό σύστημα έχει πολλά κενά και χάνονται εκατομμύρια ευρώ. Προσπαθούμε λοιπόν να οδηγήσουμε σε επιτυχία αυτή την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενίσχυση της διοικητική συνεργασίας. Αυτό είναι ένα κομμάτι του πάζλ. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους για την καλή του συνεργασία, για την καλή μας συνεργασία και πιστεύω ότι λύσεις για τα εναπομείναντα σημεία θα βρούμε αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τελευταία η κυρία Σκοτ Κέτου. Ω, δεν θα χάναμε τίποτα μια τέτοια ευκαιρία. Είναι ένα φλέγον θέμα για μένα η ΦΠΑ. Ε, όλα τα σχετικά θέματα μας τους πασίνους μας καίνε. Ναι. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ζήλε για τη δουλειά του λοιπόν. Ήμουν η για, τις βιώσιμες, ε, για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του Κοινοβουλίου και ερχόμενη από μικρή ομάδα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θεωρώ το ΦΠΑ. Επειδή ακριβώ έρχομαι από μικρή ομάδα, πρέπει να βασιστώ στη συνένεση με άλλε ομάδε του Κοινοβουλίου. Κάτι που δεν ήταν απλό, όπω φάνηκε από τι συναντήσει σκιωδών που είχαμε στο Στρασβούργο. Όπω είπε ο εισηγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το βασικό θέμα εδώ είναι η ιδέα ενό πιστοποιημένου φιλολογουμένου. Στηρίζουμε αυτή την ιδέα να ευθυγραμμιστεί το σύστημα συλλογή φόρων και να μειωθεί το διοικητικό άχθο με αυτήν την κοινοτομία. Αυτό όμω θα λειτουργήσει μόνο αν ο ορισμό του πιστοποιημένου φορολογουμένου, του φορολογουμένου προσώπου, είναι αρκετά ε, αδιαμφισβήτητο. Και θα πρέπει αυτό να συνδυαστεί και με τα άλλα θέματα, όπω ε, εκείνο τον τοσχέο που εισηγητή είναι ο κύριο Κόφοντ. Ε, βλέπουμε να υπάρχει στήριξη γενικώ προ την ε, ε, νέα έννοια του πιστοποιημένου φορολογουμένου προσώπου, ιδίω όταν υπάρχουν αμφιβολίε για παρατυπίε στην πληρωμή του ΦΠΑ. Θα πρέπει να υπάρχει κοινό έλεγχο κατόπιν αιτήματο ενό μόνο κράτου μέλου, όχι ε, δύο και πάνω. Και αυτό το στηρίζουμε. Επίση, η συμβαστική I Γιώτα. Μα ικανοποιεί για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την καταπολέμηση τη ε, φορολογική απάτη του ΦΠΑ επί τόπου. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή επιβολή των κανόνων αυτών, να θέλουμε αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε τη διασυρωριακή απάτη που ε, μα οδηγεί να χάνουμε 5 δι στα το χρόνο σε όλη την Ένωση. Και επίση να θυμίσω τι τροπολογίε μου 40 για μια αιτιολογική και 37 για το σώμα του κειμένου. Έχουν να κάνουν με τη συστηματική συλλογή δεδομένων για την φοροδιαφυγή του ΦΠΑ. Θα πρέπει ε, να συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα για να ξέρουμε πόσε ακριβώ απώλειε έχουν τα κράτη-μέλη και το μέγεθο του προβλήματο. Ελπίζω ότι και άλλε ομάδε θα στηρίξουν την ιδέα μου να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για τι κυβερνητικέ στατιστικέ και ελπίζω ότι θα ταχθούν υπέρ των δύο αυτών τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σχολιάσει για να περάσουμε και στο καθιάι και να ε, ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να συμμετέχω σε αυτήν την ε, ανταλλαγή απόψεων και όπου εξετάζεται τις τροπολογίες για την πρόταση κανονισμού για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της φοροαπάτης. Ξέρετε ότι ένα από του πυλώνε των προτάσεων που έκανε σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 για να δημιουργηθεί μια ζώνη ΦΠΑ πιο ε, σταθερή σε σχέση με τι προσπάθειε απάτη που την πλήττουν. Το Κοινοβούλιο μα έχει εξυπηρετήσει για να εγκρίνουμε όλε τι σχετικέ μεταρρυθμίσει και να πάυσουν παράτυπε προλογικέ πρακτικέ ε, καθώ και η απάτη που από ε, δυναμώνει από μια σημαντική πηγή πλούτου τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντική η ενίσχυση της δικαιωτικής συνεργασίας, ώστε οι εθνικές δικαιωτικές αρχές να μπορέσουν να αναλάβουν το ρόλο τους στην καταπολέμηση και αποδιάρθρωση των δικτύων που διαπράττουν ε, φόρο απάτη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα ε, ε, μέσα που διαθέτουμε σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό, ώστε να προστατεύονται επαρκώ οι πολίτε τη Ένωση και τα δικαιώματά του. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι ω προ την καταπολέμηση τη απάτη, ε, προτείνοντα καινοτόμε λύσει και ενισχύοντα ε, με τι ευρωπαϊκέ δράσει το δυναμικό των κρατών μελών. Η πρόταση κανονισμού αυτή Πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται πλήρως αυτές τις ανάγκες ε, και ανταποκρίνεται στην πρόκληση να δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική ζώνη. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για την πρόταση αυτή και τις τροπολογίες που προτείνατε σχετικά για να βελτιωθεί η ποιότητα του κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος για το ΚΑΤΣΤΙΑΙ? Εάν όχι, να ολοκληρώσω την εξέταση του σημείου αυτού. Ευχαριστώ τους ε, εισηγητές για την πολύ καλή συνεργασία τους που ελπίζω να επισφραγιστεί αύριο και στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν αύριο για το θέμα αυτό και φτάνουμε έτσι στο τελευταίο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης. Σημείο 7. Έλεγχος των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Πολύ σημαντικό ε, θέμα ε, αυτό που έχουμε σήμερα υπόψη, το CRR και το CRD ο κανονισμός και η οδηγία των κεφαλαιοφικών απαιτήσεων. Είναι ένας από τους γύρους ελέγχου κατά εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών μέτρων και είναι σημαντικά γιατί μπορεί να γίνουν και στο δημόσιο μέρος της συνεδρίασή μα. Μετά από τους γύρους του Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017-2018 τώρα επικεντρωνόμαστε στο CRD4 και στο CRR, τον κανονισμό και την οδηγία για τις κεφαλαιοκτικέ απαιτήσει. Ε, τα νομοθετήματα αυτά ισχύουν από το 2013 με πολλά δευτερογενή κείμενα να τα έχουν συνοδεύσει έπειτα για να βρουν ε, εφαρμογή αργότερα. Όπως θα ξέρετε, η γραμματεία της ΕΚΟΝ έχει κυκλοφορήσει κατάλογο με τα μέτρα που είναι σε εκκρεμότητα ακόμα. Θα οργανώσουμε τη συζήτηση αυτή ξεκινώντας με εισαγωγή ε, από την Γενική Διεύθυνση, μετά από την Τραπεζική Αρχή και μετά από την... Ε, τα έχουμε τις παρεμβάσεις της διαπραγματευτικής ομάδας. Ο κύριο Κάρα δεν μπορεί να είναι εδώ και ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του, αλλά θα ακούσουμε όλου του υπόλοιπου διαπραγματευτέ και μετά θα, ακούσουμε, θα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον υποδιευθυντή ε, τη Τράπεζα Υπεύθυνο για την Επίβλεψη και την Παρακολούθηση τη ε, Γενική Διεθνή ΦΥΣΜΑ. Έχετε πέντε λεπτά για την εισηγησή σα. Um, Καλημέρα. Ή μάλλον καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση, για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις, για την εφαρμογή των μέτρων επίπεδου 2, για το CRR και το CRD. Θα είμαι λογικά σύντομος. Η δουλειά για την εφαρμογή αυτών συνεχίζεται. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Είμαστε κοντά στην υιοθέτηση των τεχνικών κανονιστικών προτύπων που η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που μένουν εκρεμεί. Δεν μπορώ να σας πω ότι τα τεχνικά πρότυπα έχουν εγκριθεί πλήρως, γιατί έχουμε μια προθεσμία εξέτασης από το Μάρτιο μέχρι σήμερα που δεν υιοθετήσαμε καινούργια τεχνικά πρότυπα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάναμε και τίποτα. Δηλαδή τα έχουμε εξετάσει και έχουμε σημειώσει πρόοδο σε καθένα από αυτά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα γιατί η κατεξουσιοδότηση πράξη για το λόγο ε, κάλυψης ρευστότητας. Ε, τότε την περιασμένη φορά που σας είδα εξετάσαμε τις απαντήσεις που είχαμε λάβει για τη δημόσια διαβούλευση. Τώρα έχουμε δει όλα τα σχόλια, τα έχουμε μελετήσει, τα έχουμε διερευνήσει, έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στην κατεξουσιοδότηση πράξη μετά από αυτά τα σχόλια και τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε την ενδοϊπηρεσιακή και διαϋπηρεσιακή διαβούλευση για το εγγραφό αυτό και αν πάνε όλα καλά θα ξεκινήσουμε με την υιοθέτηση της κατεξουσιοδότησης πράξη Αυτά εν συντομία είχα να πω. Δηλαδή σημειώνεται πρόοδος, συνεχίζεται η δουλειά, συνεχίζει το διάλογος μεταξύ της δικής μας νομικής υπηρεσίας και της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Σημειώνουμε πρόοδο και σε αυτό το μέτωπο. Επομένως ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να έχουμε ε, τους επόμενους μήνες εγκρίσεις και υιοθετήσει στην πράξη όλων αυτών των τεχνικών προτύπων που είναι κρεμή. Ευχαριστώ. δεύτερος συνομιλητής μας, ο κύριος Λάρς Όβενβι. για πέντε λεπτά παρακαλώ, από το Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω. Ο Σεμπάστια να τόνισε τα σημαντικά. πράγματα και εμείς συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε διάφορους τομείς σημαντικούς για να υιοθετήσουμε τα τεχνικά πρότυπα που έχουν ήδη υποβληθεί και προταθεί. Την περασμένη φορά που σας είδα μίλησα για ορισμένα τεχνικά πρότυπα. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα είπα. Θέλω να τονίσω ότι ο αριθμός των τεχνικών προτύπων είναι ελάχιστο συγκριτικά με το, τα εκατοντάδες που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ε, καμία τα κύληση και δεν την παίρνουμε ελαφρά την καρδία. Σε ορισμένε περιπτώσει φαίνεται ότι είναι ο σωστό τρόπο. Από την περασμένη φορά έχουμε προχωρήσει ε, στη δική μας ε, ομάδα εργασίας ε, για τα πιο περίπλοκα τεχνικά πρότυπα, πώς θα εσωματώσουμε την οικονομικό κύκλο ύφεση στα μοντέλα IRB που έχουμε. Θέλουμε να κλείσουμε τις συζητήσεις μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Ουσιαστικά μας ζητήθηκε να αναγνωρίσουμε τη φύση, τη διάρκεια και τη δρυμύτητα μιας οικονομικής ύφεσης ενός αυτής της πλευράς του κύκλου. Είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα και αποφασίσαμε να διαλέξαμε να το αποσυνθέσουμε και να κάνουμε δύο έγγραφα διαβούλευσης. Το πρώτο έγγραφο διαβούλευσης, η εντολή RTS, εστιάζει στην αναγνώριση της οικονομικής ύφεση, ενώ η δεύτερη, το δεύτερο κείμενο διαβούλευσης θα συμπεριλάβει επιπρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές και περιγράφει πώς θα ενσωματώσουμε την οικονομική ύφεση που έχουμε αναγνωρίσει στη μοντελοποίηση των εκτιμήσεων. Δεν σας θα σας δώσω τεχνικές λεπτομέρειες, θα εστιάσω την προσοχή μου στο γενικότερο σκοπό. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, γιατί έχουμε μεγάλη μεταβλητότητα ε, στα αποτελέσματα που δίνουν τα μοντέλα μας από τη μία τράπεζα στην άλλη. Ακόμα και όταν έχουμε level playing field, όταν έχουμε ίσες συνθήκες και καταστάσεις για όλους. Άρα η αναγνώριση και η ταυτοποίηση ενός, ε, ε, μιας ύφεσιακής περίοδου στο πλαίσιο των μοντέλων του IRB έχει πολλαπλές διαστάσεις. Δεν, ε, εμείς υιοθετούμε μάλλον μια καθαρά μακροοικονομική προοπτική ώστε ο ορισμός μας να ε, συμπέσει με την κατανόηση που έχει κανείς ε, για την αντίληψη του τι εστί οικονομική ύφεση. Να τονίσω και το εξής. Όταν έχουμε loss given default parameters, ε, LGD δηλαδή, όταν έχουμε δηλαδή by default εξορισμού τις απώλειες να, ε, παραμέτρους σε σχέση με τις απώλειες και τις χασούρες να εντάσσονται στο σύστημα μοντελοποίησης, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε level playing field στα, στις τράπεζες. Και αυτό τονίζεται και σε κοινή επιστολή από τους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και την έχετε λάβει αυτή την επιστολή. Άρα πρέπει να έχει συνέπεια η μοντελοποίησή μας γιατί έχουμε τράπεζες με διαφορετικά δικαιοδοτικά συστήματα σε διαφορετικές χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις. Κάποιες παλεύουν να ε, κλείσουν τις απώλειες που συνδέονται, τις χασούρες δηλαδή που έχουν λόγω οικονομικής κρίσης, ενώ άλλες σε άλλες οικονομίες, άλλες τράπεζες έχουν χαμηλά επίπεδα απώλειών γιατί έχουν ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες. Και άρα ε, έχουμε ε, χαμελές επιδόσεις στο μοντέλο και χαμηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις αναλόγως. Όλα αυτά τα, όλες αυτές τις διαφορετικές συνθήκες δηλαδή και περιστάσεις πρέπει να ενσωματωθούν στα μοντέλα που χρησιμοποιούμε και στον τρόπο μοντελοποίησης για να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο με ε, αποτελεσματικό τρόπο και να είμαστε αρκετά σόφροδες και επιφυλακτικοί. Η κυρία Μπερέση για τους σοσιαλιστές παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εκ παραλλήλου να διευκρινίσω ότι το σύντομα την τελευταία φορά το θέμα αυτό, ότι σε ό,τι αφορά τι κατουσίδωτες πράξει για το ποσοστό κάλυψης ρευστότητα. θα ήταν χρήσιμο να μα πείτε γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Γιατί όταν είχε γίνει συζήτηση στο πρώτο επίπεδο ήταν ένα από τα σημεία κλειδί του κειμένου. Και το γεγονό λοιπόν αυτό, καλό θα ήταν να το λάβουμε υπόψη. Θα μπορούσατε να, λοιπόν, να μα πείτε ποιε είναι οι πρώτε πληροφορίε που έχετε να μα δώσετε από τι διαβολεύσει και στην τελική ανάλυση, αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει παρουσίαση κειμένου. Τελευταίο ζήτημα Όταν ε, δημοσιεύονται τα στοιχεία αυτά, ενώ οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, συνεχίζονται, τι γίνεται με τις εκκλησικές πράξεις τις ίδιες, γιατί η χρονική συγκυρία είναι ανησυχητική. Θα γίνει μια κινητοποίηση από πλευρά δικιά σα ή από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μενέ ε, ε, πράξει κατά εξουσιοδότηση με τη νέα νομική βάση, ενώ ουσιαστικά δεν θα έχει γίνει σταδιακή εισαγωγή και κατάργηση του προηγούμενου συστήματο. Τι θα γίνει λοιπόν, πώ θα ισχύσουν διαφορετικέ νομικές βάσει. Τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά και τη δυσκολία που αντιμετωπίσατε για την κατάσταση των απαραίτητων προτάσεων. για το νομοθετικό αυτό πακέτο. Έχετε συστάσεις να κάνετε για την λειτουργία των της πράξεων Μια και ήσασταν και εισηγητή για την αναθεώρηση των σχετικών μέτρων, θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η δική σα άποψη. Τρει ερωτήσει λοιπόν. Τι θα γίνει με πράξει κατά εξουσιοδότηση στο θέμα του συντελεστή ρευστότητα. Κατά δεύτερον, πώ θα συντονιστούμε με το επερχόμενο πακέτο και κατά τρίτον, γενικέ πληροφορίε για τη λειτουργία των πράξεων κατά σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα και τις διαβουλεύσει. Ευχαριστώ. Και μια και δεν έχουμε κανέναν άλλον στην ε, διαδικασία Catch the Eye, έχουμε μία ερώτηση, αλλά πολύ ουσιαστική. Να ρωτήσω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπέζων να μας απαντήσουν. Για να απαντήσω με τη σειρά που τέθησαν τα ερωτήματα τι γίνεται με τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Είπα στην αρχή ότι έχει σημειωθεί πρόοδο σε ό,τι αφορά τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Την προηγούμενη φορά σας ανέφερα. Είπα ότι και από τις διαβουλεύσεις και από τα κράτη-μέλη τα ίδια ακούσαμε και από τον κλάδο δηλαδή και από τα κράτη-μέλη. Εξεντήσαμε λοιπόν επισταμένως αυτά που μας είπα και προσαρμόσαμε ανάλογα το σχέδιο κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κείμενο είναι πλέον έτοιμο. Έτοιμο υπό την έννοια ότι μπορεί να περάσει στη φάση των διαθεσμικών διαβουλεύσεων. Επί της αρχής. Δεν υπάρχει και κάποιος μεγάλος λόγος για την καθυστέρηση μας πήρε κάποιο χρόνο το να διατρέξουμε τα σχόλια, να αποφασίσουμε ποια θα λεφθούν υπόψη, γιατί για να κάνω και ένα βήμα πίσω, αν θέλετε. Ο βασικός λόγος για την τροποποιητική αυτή πράξη, γιατί ουσιαστικά ήδη υπάρχει η βασική πράξη κατά εξουσιοδότηση που εγκρίθηκε το 2016 και ο στόχος λοιπόν της διορθωτικής αυτής πράξης είναι να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα τη ήδη υφιστάμενη γιατί και τα κράτη-μέλη και ο κλάδο επεσήμαναν ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τη σαφήνεια των κανόνων. Δεύτερο στόχο τώρα ήταν, σε ένα κάποιο βαθμό, να υπάρξει συντονισμός ε, των κατεξουσιοδότηση πράξεων με κάποια διεθνή πρότυπα. Αυτό λοιπόν και πράξαμε. Πολλά από τα σχόλια τα οποία απεστάλησαν στη φάση της διαβούλευσης ουσιαστικά πήγαν και πέρα από αυτό το αρχικό πεδίο εφαρμογής έγιναν προτάσεις και σχόλια τα οποία θα οδηγούσαν σε πολύ πιο θεμελιώδης τροποποίησεις της πράξης κατεξουσιοδότηση και επειδή θελήσαμε να διατηρήσουμε το όλο εγχείρημα κοντά στην αρχική μας ε, πρόταση δεν περιλάβουμε περαιτέρω τέτοια στοιχεία. Και ένας από τους λόγους που καθυστέρησε η διαδικασία ήταν ακριβώς επειδή χρειάστηκε να περιμένουμε να τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός STS για την απλή και διαφανή εξασφάλιση ασφάλειας. Γιατί έπρεπε να συμπεριληφθούν και τα στοιχεία αυτά στι καταξιοδότηση πράξη. Και δεδομένου ότι αυτό τεθεί σε εφαρμογή μόνο στα τέλη του περσινού έτου, αυτό προφανώ είχε ε, επιπτώσει στην όλη τη διαδικασία για την έγκριση τη κατεξοδότηση πράξη. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πρώτο σα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα για το πώς αυτές οι αλλαγές ε, εντάσσονται στο συνολικό πακέτο, το τραπεζικό πακέτο το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στην παρούσα φάση, δεν έχει να κάνει ουσιαστικά με τις εξουσιοδοτήσεις για Τη πράξη κατά για το ποσοστό ρευστοποίηση ε, και άρα το πακέτο όταν θα εγκριθεί δεν θα έχει επίπτωση στα LCR. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των δύο. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, κίνδυνος ε, spillover επιρροή μεταξύ των δύο σε ό,τι αφορά την έγκριση δηλαδή του τραπεζικού πακέτου. Στο τρίτο σας ερώτημα σε ό,τι αφορά η δεύτερη ερώτηση, η ερώτηση κυρία Περές, δεν ήταν μόνο για το ποσοστό ρευστότητα. όχι μόνο γι' αυτό. Μιλάμε για το σύνολο των όσων ακόμα θα πρέπει να δημοσιεύσετε. Α, συγγνώμη, έχετε δίκιο, παρανόησα. Είναι η απάντηση. Υπάρχουν φυσικά κάποιες πτυχές οι οποίες θα επηρεαστούν από το τραπεζικό πακέτο στο βαθμό που τροποποιούμε κανόνες οι οποίοι καλύπτονται στην παρούσα φάση από τεχνικά πρότυπα, ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και όχι τόσο πολύ από τις καταταξιοδότηση πράξεις, τραπεζική αρχή θα πρέπει να προτείνει κάποιες τροποποίησεις στα τεχνικά αυτά πρότυπα. Από την άποψη αυτή θα υπάρξει κάποια επιρροή και υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με την EBA σε ό,τι αφορά και το χρονοδιάγραμμα. Γιατί στο πακέτο του τραπεζικού δεν προβλέπονται νέα αμα, νέες προθεσμίες γιατί ουσιαστικά ισχύουν οι παλιέ αρχέ και η EBA πάντα έχει τη δυνατότητα να προτείνει τροποποιήσει για τα τεχνικά αυτά πρότυπα. Για πρότυπα τα οποία δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει ήδη ορίσει στο παρελθόν. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια ανανέωση των ήδη φυστάμενων ε, τεχνητών προτύπων και φυσικά το νέο τραπεζικό πακέτο εισαγάγει νέα πρότυπα, αλλά αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ο αριθμός των τροποποιήσεων που θα πρέπει να γίνουν και τα νέα τεχνικά πρότυπα τα οποία θα εφαρμοστούν θα είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με το αρχικό CRR. Και σε κάποιες περιπτώσεις οι αλλαγές των τεχνικών προτύπων θα είναι και περιορισμένες γιατί ενδεχομένω να περιλαμβάνουν μόνο περιορισμένες ε, ουσιαστικές αλλαγές. Ενδεχομένως να υπάρξει τροποποίηση υφιστάμενου τεχνητού, τεχνικού προτύπου. Άρα δεν συνεπάγεται αυτό μεγάλο γκοργασίας, αλλά και πάλι θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Αυτά σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σα Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι τώρα με την απάντηση. Τρίτο ερώτημα, τι έχουμε διδαχθεί από τον πρώτο γύρο εργασιών για τα τεχνικά πρότυπα. Νομίζω ότι έχουμε τουλάχιστον δύο σημαντικά στοιχεία να τονίσουμε καταρχάς. Να εξασφαλίσουμε ότι είναι σαφή εγκρίσει ή ευδοτήσει σε ό,τι αφορά αυτά που ζητάει και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, γιατί σε πολλέ περιπτώσει, αυτά που ζητούνται, ζητούνταν μάλλον, ήταν ασαφή. Το τι ακριβώς δηλαδή ήθελε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι δεν καλύπτονταν όλοι οι τομείς από τις αρμοδιότητες ε, τις εξουσίες όπως είχαν οριστεί. Το δεύτερο δε συμπέρασμα που εξαγάγαμε ήταν για τις προθεσμίες παράδοση σε ό,τι αφορά τα τεχνικά πρότυπα. Σε κάποιες περιπτώσεις ήμασταν υπερβολικά αισιοδόξοι. Υπερβολικά αισιοδόξοι γιατί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τεχνικά πρότυπα για πολύ περίπλοκα τεχνικά ζητήματα και πολύ ευρεία ζητήματα, όπω για παράδειγμα οι μεθοδολογίες αξιολόγηση των μοντέλων, πήραν πολύ παραπάνω χρόνο από ό,τι αρχικά πιστεύαμε, γιατί τα θέματα αυτά ήταν τεχνικά στη φύση τους και ευρύτατα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δώσουμε πιο πολύ προσοχή στα πρότυπα για τεχνικά αυτά ζητήματα. στις προστασμίες και τεχνικά πρότυπα από, τις, ε, από την παραχώρηση αρμοδιτήτων και εξουσιών πάνω από 100 σε αριθμό. Θεωρώ ότι στα πιο περίπλοκα ζητήματα ε, υπήρχε κάποια καθυστέρηση, αλλά γενικά η διαδικασία λειτουργήσε σωστά. Φυσικά είχαμε κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα στην αρχή. Γιατί και εμείς οι ίδιοι έπρεπε να εξοικειωθούμε με τη διαδικασία. Τώρα νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών πάει μια χαρά. Θα πάμε πολύ καλύτερα από ότι στην αρχή. Φυσικά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση και στην εργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή, Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για να βελτιστοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία στο βάθμο το δυνατό. και σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες. Κάτι που πάντα ξεχνάμε να συνυπολογίσουμε είναι ότι αυτά τα πράγματα κινούνται κάπως σε κύματα. Και δεν είμαστε εκεί μοναδική μονάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συχνά συμβαίνει για παράδειγμα και η νομική υπηρεσία και η μεταφραστική υπηρεσία έχουν και άλλες ασχολίες. Δεν έχουν μόνο εμάς στο κεφάλι τους. Και όλα αυτά είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν ε, ορίζουμε τις προθεσμίες για τα τεχνικά πρότυπα. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ναι, να θίξω κι εγώ τα ίδια με αυτά που είπε ο Σεμπάστιαν. υπάρχουν παράπλευρες συνέπειες, όπως οι εκθέσεις για τη ρευστότητα. Θα χρειαστεί χρόνος. Και χρόνος μπορεί να δοθεί και στις εταιρείες για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Για την αλληλεπίδραση για τα τεχνικά πρότυπα των τραπεζών το πρόβλημα είναι ότι κάποιε φορέ υπήρχαν καθυστερήσει λόγω τη δέσμη μέτρων για τι τράπεζε που υπήρχαν ταυτόχρονα. Ο κίνδυνο είναι ότι πρώτα θα έχουμε σχεδιασμό των τεχνικών προτύπων, θα, ισχύ, θα ισχύσουν για λίγο καιρό και μετά ε, βάσει των υπόλοιπων που συζητιούνται από τους πολιτικούς ευθύνοντες μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Λόγω χάρη ο κύκλους ύφεση. Με τη Βασιλεία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Τη συζητήσαμε πολύ τη Βασιλεία, αλλά τελικά δεν υπήρξε κάτι τόσο συμπερασματικό σε αυτό το τομέα. Οπότε πρέπει να λάβουμε διαφορετικά μέτρα μετά. Τα διδάγματα που αντλήσαμε εδώ, ήδη πολύ παρόμοια με αυτά που είπε ο Σεμπάστιαν, βλέπουμε ότι οι χρονικές γραμμές της τραπεζικής αρχής δείχνουν μεγάλο βαθμό φιλοδοξία από πλευρά της CBA. Ιδίω στο τεχνικό σκέλος για το τι θέλουμε να πετύχουμε. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 12 μήνε για τα σωστά τεχνικά πρότυπα. Τρει ε, μήνες διαβουλεύσεις, ε, οι διαδικασίες λήψης απόφασης και ούτω καθεξής. Τουλάχιστον ένα χρόνο. Και για τη νέα πρόταση, την ε, οδηγία για τις κεφαλικές απαιτήσει νούμερο 2. Πάλι θα χρειαστούν 6 μήνες τουλάχιστον. Είναι μη ρεαλιστικό ότι θα προλάβουμε όλα βάσει τις εμπειρίες μας. Και για μερικά από τα ζητήματα με την ε, νομική μας εντολή. Με τα τεχνικά πρότυπα δεν μπορούσαμε να απειλήσουμε όλα τα ζητήματα, διότι υπάρχουν ε, περιορισμοί για το πώ έχει σχεδιαστεί η εντολή. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με τι νομικέ υπηρεσίε τη Επιτροπή που έχουν τη σχετική ερμηνεία. Και αυτό είναι ένα τομέα όπου θα θέλαμε μια επίσημη ευκαιρία να εξεταστεί η εντολή που έχουν αποφασίσει οι νομοθέτε βάσει του τρεμερού διαλόγου. Και να δούμε τα πράγματα από μια σκοπιά λίγο πιο τεχνική. Θα ήταν πολύ χρήσιμο και για τις δύο πλευρές αυτό για να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα επιπλέον προβλήματα που είχαμε στη διαδικασία υλοποίηση. Όπω είπε και ο Σεμπάστιαν, η διαδικασία αυτή από πλευρά μα είναι εν εξελίξη. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή για να εγκριθούν και τα υπόλοιπα τεχνικά πρότυπα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπερές θέλει επερώτηση. Ναι, μια ακόμα ερώτηση. Γιατί είπατε ότι θα υπάρχει επικάλυψη μεταξύ της συνεχιζόμενης δουλειάς και την αναβολή της διαδικασίας περιμένοντας το νέο πακέτο να έρθει επιτάπητος. Ελπίζω ότι έχετε σαφώς εντοπίσει ποια είναι τα τεχνικά πρότυπα που θα τα αφορά η αλλαγή. Θα ενημερώσετε το Κοινοβούλιο για την αλλαγή ή θα τα μάθουμε όταν προκύψουν οι αλλαγέ. Διότι αν έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση επειδή περιμένετε το πακέτο για τι τράπεζε, δίκαιο θα ήταν το κοινοβούλιο να το γνωρίζει. Ευχαριστώ, παρακαλώ, πολύ σύντομα. Νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις αποστέλουμε επιστολή στην αρμόδια επιτροπή. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον. Ε, και αναφέρουμε και το Κοινοβούλιο ε, αυτά τα δημοσιεύουμε στον ιστοτοπό μας. Ευχαριστώ να σα δώσω το κατάλληλο link. Όποτε υπάρχουν καθυστερήσεις, ε, δημοσιοποιούμε τα σχετικά στοιχεία. Προσπαθήσαμε να είμαστε σαφείς στην επικοινωνία μας και να το καταστήσουμε και δημόσιο. Εάν κάτι από αυτά δεν έχει πάει καλά, ευχαριστώ να το κοιτάξω εάν μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας. Όμως σε κάθε περίπτωση έχουμε ενημερώσει για τις συγκεκριμένε δυσκολίες και εσωτερικά χωλήματα. Ευχαριστώ. Ε, φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές, τους προσκεκλημένους μας και να κηρύξω τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Αρχίζουμε αύριο στις 9 το πρωί με την ακρόαση του Γενικού Γραμματέα του ΩΣΑ. Καλό σας βράδυ κάπως μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε προβλέψει. Ευχαριστώ.